we start there. You can. Well, if I can uh, start and. Uh, Επιτρέψτε μου να αρχίσω, λέει ο Πρόεδρο. Να συνεχίσουμε τι εργασίε μα. Έχουμε τώρα. Το θέμα μας είναι Ορισμένα μέτρα κατά το χρόνο που επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμη αλληλεία με στόχο διατήρηση των αποθεμάτων. Συγχαρητήρια, ο κύριος ε, Πόγκα, Επιτροπή Αλία. Επαναλαμβάνει ο πρόεδρο. Διεξαγωγή μη βιώσιμη αλίας για διατήρηση αποθεμάτων. Είναι, πρόκειται για την πρώτη ανάγνωση. Κύριε Πόγκα, έχετε το λόγο. Merci, Monsieur le Président. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δύο λόγια να σας πω. το έγγραφο αυτό το οποίο έχουμε προετοιμάσει για την Επιτροπή Αλίας, για αυτά τα μέτρα. Οι χώρες που επιτρέπουν την εξαγωγή μη βιώσιμης αλίας. Ο στόχος είναι η διατήρηση των ηχθειαποθεμάτων. αποθεμάτων. Πρώτα πρώτα. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο κανονισμού. Εκεί έχουμε μια νέα μεταπολιτική για κάποια βιώσιμη αλία, η οποία να χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα παντού σε όλο τον κόσμο. Επίση, ε, εδώ ε, έχουμε ε, παραπομπή στον για την παρανομή αλία, την αλία που δεν περνάει από κάποια ρύθμιση. Ε, πάρα πολύ ε, σωστό ήταν το, το, το, το, θέμα το οποίο ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έτσι έχει ε, ένα πάρα πολύ σημαντικό όπλο για αυτούς τους σκοπούς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα-πρώτα, σας υπενθυμίζω ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να έχουν μια διαφορετική μεταχείριση και να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική, η διοικητική και η οικονομική του κατάσταση. Επίση, τα μέτρα αυτά τα οποία θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διέπονται από κάποια συνέπεια σε σχέση με τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε ε, για την ανάπτυξη. Και σα παραπέμπω τώρα στην ιδεολογική παράγραφο 5 και στο άρθρο 5 ε, και το άρθρο 4 του κανονισμού. Επίσης έχουμε εδώ τώρα μια ρήτρα Παρακολούθηση και ελέγχου, ούτω ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα να ενημερώνεται για την εφαρμογή του κανονισμού και να τον προσαρμόσει ανάλογα. Γι' αυτό και εγώ εδώ έχω προσθέσει ένα καινούριο άρθρο, το άρθρο 8α. Νέο άρθρο. Αυτά, Πρόεδρε. Είμαι στη διάθεσή σα για οτιδήποτε ε, παρατηρήσει. Η δε προθεσμία για τι τροπολογίε είναι η 7η Μαρτίου το μεσημέρι και σας ευχαριστώ. Η Ζαμπέλα που είναι η σκιώδη συγγύτρια ασχολείται με άλλα θέματα λύση και δεν μπορείς να παραστεί σήμερα. Πάντως, η θέση μας και η θέση της είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα προσεκτικοί όσον αφορά τις εξαιρέσεις, παρεκκλήσεις για τα θέματα της μη βιώσιμης αλίας. Διότι τελικά είναι ύψος της κάθε χώρας να, να μπορέσει να διατηρήσει τους ελεύθερους πόρους γιατί θα υπάρχουν ψάρια αλλιώς. Οπότε προσοχή, προσοχή στις εξαιρέσεις από μια τέτοια αντιμετώπιση. Βεβαίω και θέλουμε να έχουμε κάποιε διατάξει, ούτω ώστε οι αντισόμενε χώρε να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαχείριση τη ε, αλληλεία γενικά, τη συμμετοχή του σε κάποιου φορεί που ρυθμίζουν τι ε, διαφορέ και είπαμε ότι θα πρέπει να, ρυθμίσουμε τις ε, προϋποθέσεις που βοηθούν για τη, βιώσιμη αλληλεία, να δούμε τι θα γίνει με, αυτές, αυτό το είδο τι πρακτικέ που παραβλάπτουν ε, με, με κάποιο είδος βιομηχανική αλληλεία, με σχετικέ εγκρίσεις που δίνουν οι αντιμετωπιστές χώρες, οπότε να μην έχει παραθυράκια ο νόμος, ούτως ώστε οι χώρες που αλλιεύουν να μπορούν με αυτά τα παραθυράκια να εκμεταλλευτούν την προτιμησιακή μεταχείριση των εξωμένων χώρων. Επίσης, οι κυβερνήσει ε, των χωρών αυτών θα πρέπει ε, να είναι υπεύθυνε για αυτά τα οποία κάνουν και επίσης να υπάρχει διαφάνεια σε σχέση με τις ε, αλληλευτικές άδειες που εκδίδονται. Άρα θα πρέπει να είναι συνεπής πως μια τέτοια ε, πολιτική βοηθάει τη βιώσιμη αλληλεία για να ε, τηρούν επίση τι διεθνεί συμφωνίες. Θα πρέπει επομένω το ρυθμιστικό πλαίσιο να ενδυναμωθεί, ε, υποδομές, όπως τα λέει εδώ η έκθεση με το οποίο συμφωνούμε επίση, Να δούμε τι γίνεται όσον αφορά του, αυτούς που αλλιεύουν σε μικρή κλίμακα και που ψαρεύουν για εσωτερική κατανάλωση. Άρα, άρα, γι' αυτό σας λέω, όσον αφορά την βιώσιμη αλία, προσοχή, προσοχή στις εξαιρέσεις. Η Ιζαμπέλ ε, θα είναι στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε. Πρόεδρος. Ο κύριος Λέβεν. Κυρία Λέβεν, τέλος πάντων, μας τα είπε χθες όσον αφορά ε, τις χώρες αυτές οι οποίες θέλουμε να βοηθήσουμε όσον αφορά τους αριθμούς πόρους που διαθέτουν και όπου και εμείς ψαρεύουμε. Άρα, ακούσαμε την κυρία Κέλλερ, θα τα λάβει αυτά υπόψη ο κύριος Πόγκα και να εντάξουμε αυτές τις αρχές που μας εξηγήθηκαν στο σώμα της εκθέσης. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Όχι, Δηλώ, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Πόγκα, για το έγγραφό του, την έκθεσή του. Διαπιστώνουμε με χαρά μας ότι συμφωνεί και ο Σπόγκα με τις θέσεις μας. Βεβαίω και είναι θεμητές οι ανησυχίες του όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και εμείς στο κείμενό μας έχουμε θίξει το ζήτημα αυτό. Για μας είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να κατοχυρωθούν τα συγκεκριμένα συμφέροντα των χωρών εκείνων. Όσον αφορά τώρα την ρήτρα αναθεώρησης, Ξέρετε ότι έχουμε αλλεργία σε τέτοιου ρήτρε καταρχήν. Πάντω μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια χωρί να έχει ακόμα αρχίσει να εφαρμόζεται ο κανονισμό αυτό. Και αν στην περίοδο αυτή χρειαστεί. Θα δούμε, γιατί ακριβώ και στο παρελθόν παρόμοιε ρυθμίσει δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα. Είναι αρμοδιότητα και υποχρέωσή μας να είναι ενεργός ο κανονισμός και όταν θεωρηθεί απαραίτητο να προβαίνουμε στην αναθεωρησή του. Ευχαριστώ. Thank you. Um, anybody else? Ευχαριστώ. Θα ήθελε κάποιος άλλος τον λόγο. Όχι, όπως είπαμε λοιπόν η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Α, όχι, ο ίδιος ο κύριος Πονγκά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε σχέση με τις ε, εξαιρέσεις και παρεκκλήσεις οι οποίες εγκρίνονται στις συμφωνίες. Ε, υπογραμμίζω αυτό που είπε η Επιτροπή για την αναθεώρηση του κανονισμού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί αν πράγματι υπάρχουν λάθη και από τις δύο άλλωστε πλευρές, καλό θα είναι να επανέλθουμε στο σωστό δρόμο. Θα λάβω υπόψη μου λοιπόν τις παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν για το επόμενο στάδιο. Ευχαριστώ κύριε Πόγκα. Είπαμε λοιπόν 12η Μεσημβρινή 7η Μαρτίου προθεσμία κατάθεση των απολογιών. Ψηφοφορία θα γίνει την 27η Μαρτίου. Περνάμε στο επόμενο θέμα, σημαντικό και αυτό. Νέα αναπτυξιακή συνεργασία με τη Λατινική Αμερική. Ο κύριος Λάστρα έχει το λόγο οι χώρες της Λατινικής Αμερικής ε, ε, ενισχύουν την ολοκλήρωσή τους από τις δεκαετίες του 70 και μετά. Εμείς δεν είμαστε μόνο σημαντικός εταίρος εμπορικός, αλλά είμαστε και ο δεύτερος πιο σημαντικός δωρητής στην περιοχή. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν. Πρέπει η Επιτροπή μας να λάβει υπόψη τις αλλαγές στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσουν σύντομα. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τίνει στη μείωση ε, της στήριξης προς τις χώρες μεσαίου ε, εισοδήματος και η περιοχή αυτή ακριβώς βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Η Βραζιλία θα γνωρίζετε ότι τον προηγούμενο μήνα ξεπέρασε την Μεγάλη Βρετανία σαν η έκτη μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη στον κόσμο. Πρέπει λοιπόν η παρέμβασή μας να συνεχίσει ε, να βοηθά τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ε, ιδιαίτερα στον τομέα της ανάπτυξης. Ιστορικά η Αργεντινή στη, στο, στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν η τρίτη πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. Βέβαια έχουν ε, αλλάξει πολλά από τότε, αλλά νομίζω ότι το θέμα που μας απασχολεί έχει και μία διάσταση σε σχέση με τη σταθερότητα της περιοχής και δίνω το λόγο στον κύριο Λάστρα. muchas gracias, presidente. Eh, ε, en primer lugar, ε, Πρώτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους με όσους έχω συνεργαστεί γιατί χρειάστηκε για το σχέδιο αυτό εντατική δουλειά. Ευχαριστήσω και όλες τις μη οργανώσεις που από την πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα μου για να διαμορφώσω αυτό το κείμενο επίσης για την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την ΔΕΦΚΟ, τους εμπειρογνώμους για την ε, Λατινική Αμερική και ε, βεβαίως τον ΟΗΕ. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνούμε, επομένως, τη συμβολή όλων αυτών για τους οποίους και πάλι ευχαριστώ. Τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι αξίζει να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με αυτά τα θέματα. Μεταξύ λοιπόν το 90 και 2010 κατά 17 μονάδες μειώθηκε η φτώχεια και είναι 12,3% τώρα το ποσοστό ε, αυτών των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια στην Νότια Αμερική. Από την άλλη μεριά πρέπει να διαπιστώσουμε ότι θα πρέπει να δούμε αυτά τα στοιχεία. Ε, είναι τέτοια που μας προβληματίζουν γιατί συνεχίζονται αυτά τα προβλήματα στην Νότια Αμερική. Έχουμε 73 εκατομμύρια ακόμη Νότιο-Αμερικανών οι οποίοι ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Μέσω αυτής της ΤΕΠΑΛ 10 από τις 15, 10 από τις 15 χώρες που βρίσκονται στην κατάσταση βρίσκονται στην Νότια Αμερική. Όλα αυτά επομένως είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Επομένως θα πρέπει οι χώρες οι σχετικές να, να θεωρήσουν τις, ε, την πολιτική τους και να βοηθήσουν στο να καταπολεμηθεί η φτώχεια σε αυτή την ε, περιοχή. Να δούμε επομένως με τι μέσα πολιτικής θα μπορέσουμε να κρυβώσουμε τη φτώχεια πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην ξεχνούμε, όπω είπαμε προηγουμένω, ότι έχουμε αυτά τα 180 εκατομμύρια που συνεχίζουν να χρειάζονται τη βοήθειά μα. Οπότε και εμεί, επομένω, γι' αυτό και είμαστε ο πρώτο εμπορικό εταίρο, βασικό δωρητή. Οπότε η αρρωγή που αυτά τα χρόνια δίνουμε μέσω διαφόρων συμφωνιών και των συμφωνιών σύνδεση και κυρίω αναπτυξιακή ε, αρρωγή, όλα βοηθήσαμε να βοηθηθεί και η κατάσταση. Το 2012 θα, κατά τρεις ή τέσσερις μονάδες θα αυξηθεί η ανάπτυξη. Βέβαια κάποιες άλλες χώρες όπως το Μεξικό και η Κεντρική Αμερική έχουν χτυπηθεί από την ε, παγκόσμια κρίση. Επομένως, συνεχίζει διαπιστώνει το δυνατό ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτη η Λατινική Αμερική ε, υπό τη σημερινή συγκυρία της κρίσης. Επομένως, θα πρέπει να συνεχίσουμε τη βοηθειά μας και να δούμε την προστιθέμενη αξία την οποία έχει ανάλογα με τις ε, ειδικέ ανάγκες που έχει κάθε χώρα και κυρίως ανάλογα με το μέσο εισόδημα, ούτως ώστε να βοηθήσουμε να έχουμε λιγότερες ανισότητες, να καταπολεμήσουμε την ε, τη φτώχεια και να προχωρήσουν οι περιοχή στην ανάπτυξη. Άρα θα πρέπει να συσφίξουμε τις ε, σχέσεις με τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε στην άκρη που είναι Αμερική, δεν είναι δυνατόν να δούμε την εντύπωση ότι δεν αποδίδουν τη σημασία που έχει αυτή η περιοχή πέραν ε, των δεδομένων εμπορικών και λοιπά σχέσεων. Άρα Αντίστοιχε είναι και οι προτάσει που κάνουμε με αυτό το κείμενο και πάρα πολλέ χώρε τη Νοτιοαμερική θέλουν να μην είναι απλώ αποδέκτε βοηθεία, αλλά θέλουν να μπουν σε μια καινούργια δυναμική μορφή συνεργασία. Κατά τον τρόπο, επομένω, θα πρέπει να βοηθήσουμε τι χώρε με τρόπο αποτελεσματικό. Δεν συμφωνούμε με τις πρώτες Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χρησιμοποιεί αποκλειστικά σχεδόν οικονομικά κριτήρια Εκουαδόρ, Κολομβία έτσι θα, θα βγουν από το πλαίσιο βοηθείας. Θέλουμε να υπάρχει διαφοροποίηση στην ε, αρρωγή, αλλά να είναι με υπεύθυνο τρόπο. Τα κριτήρια δεν ε, λαμβάνουν υπόψη το πόσο είναι μια χώρα και έχουμε κάποιους άλλους νέους δείκτες, νέα κριτήρια και άρα η διαφοροποίηση να γίνεται στην φάση του προγραμματισμού και κατά αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και επομένως κατά αυτόν τον τρόπο να στείλουμε το σωστό μήνυμα στους νοτιοαμερικανούς εταίρους μας. Ε, και άλλες περικοπές προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάνε σε θεματικά προγράμματα κάποια χρήματα τα οποία θα φύγουν από χώρες οι οποίες έχουν λιγότερη, ε, λιγότερη ανάγκη. Οπότε θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις, τη βοήθειά μας στους πιο ευάλωτους και άρα έτσι να βελτιωθεί η νοτισιακή βοήθεια. Το, το, το DCI 2014 μέχρι το 2014 θα πρέπει να υποστεί μια καινούργια κατανομή των πόρων ούτω ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε για την εγκρίζωση της φτώχειας στις χώρες που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Επίσης, η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής κόβει εντικά χώρες από την συνεργασία. Ούτε με αυτό συμφωνούμε. Άρα θέλω να γίνει καινούριο προσανατολισμός του, του DCI. Να μην έχουμε περικοπέ, μην έχουμε διακοπή τη διμερούς συνεργασία. Άρα να βρούμε τις, ε, τους τρόπους που είναι οι πιο καλά προσαρμοσμένοι στις αυτών των χωρών. Κολομβία, σημερινό και Περού να συνεχίσουν να καλύπτονται. Και μόνο έτσι να έχουμε μια συνεπή στρατηγική. Και να είναι μόνο βαθμία η προσαρμογή της α, ε, διμερούς βοηθείας συνεργασία, προγράμματα τα οποία να συνεχίσουν να είναι ενεργά και να έχουμε μια μεταβατική περίοδο για την ε, συνέχιση της διμερούς συνεργασίας. Τέσσερα χρόνια είναι αυτή η μεταβατική περίοδος. Επίσης, Ε, η πρικοδότηση επίσης είναι ε, συμπληρωθεί με ένα δις για τις χώρες με μέσο εισόδημα. Βάσει του κανονισμού δεν μπόρεσα να περιλάβω και άλλες προτάσεις που θα ήθελα σε αυτό το σχέδιο Όλοι επομένω ελπίζω ότι θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση του κειμένου με τροπολογίε, όλε οι πολιτικέ πτέρυγες. Έχω και εγώ ήδη κάπου 20 τροπολογίε για να δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία, την κοινωνική συνοχή, την συνεργασία βορρά-νότου, την καταπολέμηση τη εγκληματικότητα, την υγεία, την παιδεία, την αλλαγή του κλίματο, την ε, τεχνολογική συνεργασία και επίση θα πρέπει να έχουμε ακόμα συνεπέστερη πολιτική για την ανάπτυξη. Τώρα, οι τροπολογίε ε, θα πάμε στην καλύτερη κατανομή ε, των, πόρων στην περιοχή. Ε, δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε περισσότερη κοινωνική πρόνοια και επίσης φορολογική αντίστοιχη πολιτική. Επίσης κάτι για την, για την παιδεία, γιατί είπαμε ότι τώρα υπάρχει, υπάρχουν μεγάλε ανισότητε στο σύστημα παιδείας τη περιοχή. Επίσης, να βελτιωθεί η πρόσβαση των, των φτωχότερων στην παιδεία και στη, στην ε, κατανομή του πλούτου καινοτομία, τεχνολογία και επίσης να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η παραοικονομία εμποδίζει την ε, κοινωνική κινητικότητα. Κυριαρχεί η παραοικονομία. Έχουμε μεγάλες μισθολογικές ανισότητες. Δεν προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Ούτε έχουν ιατρική κάλυψη. Έτσι επομένως να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές κατά τις φτώχειες των ανισοτήτων με πολιτικές που θα εγγυώνται την απασχόληση και νομισματικά μέτρα τα οποία και αυτά να κατατείνουν στη βοήθεια των μη προνομιούχων. Επίσης έχουμε προγράμματα ε, διάφορα για την παιδεία ούτω ώστε το ευρωλάκι είναι ένα ίδρυμα το οποίο είναι πολύ δυνατό, το οποίο πρέπει να, να εκμεταλλευτούμε. Επίση, κοινέ προτάσει για την ε, οικονομία, την παγκόσμια, για, το, για την αλλαγή του κλίματος, ε, να, μπορούμε μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε πάνω έτσι με την Λατινική Αμερική τι καινούργιε προκλήσει. Να μην ξεχνούμε για τα καινούργια τη η ΕΕ κάποια βασικά θέματα οπω τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιση να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστεί η βία κατά των ε, γενικών και επίση τα θέματα σεξουαλική υγεία. Επομένω περιμένω πώς και πώς να ακούσω τι παρατηρήσει σα και να λάβω υπόψη ότι θα πείτε και να συνεργαστείτε όσο γίνεται πιο δυναμικά στην επεξεργασία αυτή τη ε, έκθεση που πρέπει πραγματικά να αντικατοπτρεί τι απόψει τη Επιτροπή μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρον τα τόξα μα είπατε, ιδιαίτερα το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αγνοήσει ή τέλος πάντων παραγνωρίσει τη Λατινική Αμερική στο παρελθόν. ότι έγιναν κάποιε προσπάθειε, αλλά τα αποτελέσματα ισχνά. Αυτό που πράττουμε τώρα φαίνεται πολύ πιο σημαντικό για τον κόσμο στη Λατινική Αμερική. Θέλουμε να κάνουμε κάτι καινούριο και ανάλογα με την Ασία, όπου έχουμε πολύ μεγάλες ε, μεγάλους θύλακες φτώχειας. Στη δε Λατινική Αμερική που δεν γνωρίζει καμία χώρα μικρού εισοδήματος, κάτω του εισοδήματος, αλλά μόνο μία ε, μεσαίου εισοδήματος, lower income δηλαδή, την Ικαράγουα, ε, είναι επίσης πολύ σημαντικό να δραστηριοποιηθούμε. Κυρία Κέλλερ, ναι και εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο για την έκθεση, συμφωνούμε απολύτως, ιδιαίτερος μας ικανοποιεί η έμφαση που δίνεται στο γεγονός ότι η μεταρρύθμιση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε υποχρέωση για τις χώρες αυτές να υπογράψουν, να κυρώσουν συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Γενικά η προσέγγιση σας προς τις λατινοαμερικανικές χώρες και η υπογράμμιση της ε, ανάγκης να ε, στηριχθούν άλλα κριτήρια και όχι μόνο τα DNA της Παγκόσμιας Τράπεζας στην οποία αναφέρεστε μας ικανοποιεί ιδιαίτερως. Επίσης, η πολέμηση της φτώχειας έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, συμφωνούμε απολύτως, και αναφέρεστε σε τροπολογίες που περιμένετε να δείτε εμείς μάλλον για να συμπληρώσουμε παρά για να αντικαταστήσουμε κάτι, θα καταθέσουμε τροπολογίες. πίν στην ε, κοινωνική συνοχή, ε, την οποία αναφέρατε και εσείς ασφαλώς και θα συμφωνήσουμε. Κάποια σημεία θα ήταν ενδιαφέροντα για τροπολογίες. Είναι και όπου ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πόροι τυρισμένοι για την ανάπτυξη στην Λατινική Αμερική να μην αποβούν τελικά εις όφελος άλλων δραστηριότητων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ασφάλεια, ενέργεια ή εμπόριο και επίσης ότι θα πρέπει να υποστηρίζονται οι μεγάλες ε, κλίμακας ε, παραγωγές ε, βιοκαυσιγεωργικών καυσίμων. Επίσης αναφέρεστε στο μέσο επενδύσεων για τη Λατινική Αμερική όπου πιστεύουμε πως θα πρέπει να υπογραμμιστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των δαπανών για τις μεγάλες υποδομές. Όλο και πιο πολλά χρήματα δηλαδή θα δαπανώνται για μεγάλες υποδομές, αλλά χωρίς καμία διαβούλευση με τους τοπικούς πληθυσμούς και χωρίς καμιά ε, μέρημνα για τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να το σημειώσουμε, το είπαμε και χθε. Και επίσης μια τροπολογία θα μπορούσε να αναφέρεται στην συμμετοχή και στι διαβουλεύσεις των μέσων για την ε, Λατινική Αμερική ώστε να ε, παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και τη συνεργασία των με αυτόν. Αυτά. Ίσως θα μπορούσαμε να αναφερθούμε όμως και σε μια συμπληρωματικά, σε μια δυνατότητα για, για συνεργασία με την, ε, στον τομέα της δικαιοσύνης με τις Λατινοαμερικανικές χώρες ή στην καταπολέμηση της ατιμορρησίας που ασφαλώς γνωρίζετε καλύτερα από μένα ως ζήτημα. Ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί σχέση με τις λατινοαμερικανικές χώρες. Πάντως ευχαριστώ. Είμαστε εν γέννη ικανοποιημένοι με την έκθεσή σας και ε, μπορούμε να βρούμε, πιστεύω, μια ε, συμφωνία ως προς τροπολογίε. Κύριος Φυσάς Αοξέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρούμε τον κύριο Λάστρα, διότι είναι υπέροχο το σχέδιο εκθέσεως το οποίο συνέταξε. Στι γενικέ ε, γραμμές ε, συμφωνούμε με το κείμενο αυτό. Οπότε όπως πάντα θα συνεργαστούμε πάρα πολύ σωστά για να κάνουμε ε, να, να, βάλουμε τις πινελιές που χρειάζεται ούτως ώστε να δούμε ε, πώς θα βελτιώσουμε το κείμενο. Μια που είπαμε ότι επί της ουσίας του, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το κείμενο. Ε, ε, εξορισμού υπάρχουν περιορισμοί στη σύνταξη κάποιας έκθεσης. Άρα οποιαδήποτε έκθεση επιδέχεται βελτίωση με τις τροπολογίες. Επίσης θα ήθελα να σας πω δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα τώρα να προβούμε σε περικοπές στην ε, ε, βοήθεια προς την Λατινική Αμερική. Γιατί στο συγκυρία αυτή της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης οι χώρες Λατινικής Αμερικής τα πάνε καλά σχετικά με το τι υφιστάμεθε εδώ στην Ευρώπη. Όμως, παρόλα αυτά, παρόλα αυτά η κρίση τους επηρεάζει αρνητικά. Αν όμως εμείς τους κόψουμε από τη βοήθεια, και τότε θα πλήξουμε την, τις, τις καλές σχετικά επιδόσεις που έχουν τώρα. Άρα τώρα είναι η λάθος στιγμή να προβούμε σε περικοπές. Τώρα, θέλω και εγώ να σταθώ σε κάποια σημεία τα οποία μου φαίνονται σημαντικά. Η ανασφάλεια που πριν ανέβει σε αυτές τις χώρες, γιατί πολλά από αυτά τα, ε, τα, τα, τα, τα κράτη πρέπει να ξεδεύσουν πολλά λεφτά ε, για θέματα ασφάλειας, άρα, άρα, άρα, άρα εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Είναι πολύ σημαντικό. Και εάν αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, τότε αυτές οι χώρε θα έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα. Άρα, τα χρήματα τα οποία διαθέτουν τώρα για τα θέματα ασφάλειας θα πάνε σε αναπτυξιακή πολιτική. Και οι χώρε αυτέ θα καταστούν ακόμα πιο ελκυστικέ αγορέ. Για τη φτώχεια τώρα. Ε, υπάρχουν ε, πολλές και μεγάλες ανισότητες μεταξύ των χωρών αλλά και μέσα σε κάθε χώρα. Ένας στους τρεις Νοτιοαμερικανούς ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Και όπως είπαμε 10 ε, από τις λατινοαμερικές χώρες είναι μεταξύ των 15 πιο άνισων οικονομιών στον κόσμο. Άρα η ανακατανομή του πλούτου θα πρέπει να γίνει με δίκαιο τρόπο, δικαιότερο τρόπο τόσο ώστε να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Άρα και αντίστοιχα πρέπει να δική μας συμβολή. Και γι' αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουμε την ενίσχυση σε παιδεία, υγεία, καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος και επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ. Ε, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το πώς έτσι θα βοηθηθεί η ανάπτυξη μέσω των ΜΜΕ και άρα γι' αυτό και θέλουμε συγκεκριμένα προγράμματα όπως τα λέει και η έκθεση. Ίσως μπορούμε και να επεκταθούμε. Ε, να βοηθούν οι γυναίκες, επιχειρηματίες και να τονωθούν οι επενδύσεις. Επίσης, να δούμε το θέμα και λίγο εγωιστικά ούτως ή από Ευρώπης δηλαδή Έχουμε κάποιες ε, χώρες που είναι πιο πλούσιες, πιο, πιο, πιο υψηλό βιωτικό επίπεδο να αποκτήσουν οι χώρες της Νοτιοαμερικής. Αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε καλύτερη αγορά να κατευθυνθούμε εμείς. Άρα μας συμφέρει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση και έτσι να μπορούμε να πουλήσουμε καλύτερα τα προϊόντα μας. Ακριβώς επειδή τώρα σοβεί η κρίση. Δεν θα είναι θετικό να ανακοπεί αυτή η θετική οικονομική πορεία των χωρών εκείνων. Θα ήταν επίσης αντιφατικό να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια σε κάποιες χώρες όπως η Αφρικανική Δημοκρατία και από την άλλη μεριά να κόβουμε τη βοήθεια στο Περού, στον Ισημερινό, την Κολομβία. θα έπρεπε ομένως να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά για χώρες συγκρίσιμες. Ο κύριος Ντεμέρα. Εγώ, Πρόεδρε, θέλω να σχολιάσω με τη σειρά μου την έκθεση Κορτές και τόσο είπαν και οι συνάδελφοι, διότι σε γενικέ γραμμές συμφωνώ με την έκθεση του Ρικάρντο. Επίσης, συμφωνώ με τις τροπολογίες του, με τις ε, προθέσεις του, με εξαίρεση το τελευταίο το οποίο ανέφερε. Γενικά νομίζω ότι θα σημειωθεί συνένεση μεταξύ των μεγαλύτερων πολιτικών πτερίγων του Κοινοβουλίου. Αυτό με το οποίο διαφωνώ είναι τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι δεν είναι ρεαλιστικά. Α, ε, αγνοούν την λατινοαμερικανική πραγματικότητα. Πολύ σωστά αυτά τα οποία είπε ο προλαλής σας, ο κύριος Φίσας για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με την Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία και κάποιες λατινοαμερικανικές χώρες. Φυσικά και πρέπει κάτι να γίνει για την ασφάλεια και την ανασφάλεια, όπως τα είπαμε. Να βοηθήσουμε για παιδεία, υγεία, υδροδότηση, ενέργεια. Αλλά θα πρέπει να δούμε επίση τις συνέπειες της ε, ανασφάλειας για την Ευρώπη. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοια προβλήματα σε πάρα πολλές χώρες στην Νότια Αμερική. Ναρκωτικά, δεδομένο έγκλημα. Και έχουν διαβρώσει τους θεσμούς, τα θεσμικά όργανα, την κοινωνία των πολιτών, τη δικαιοσύνη, την αστυνομία, την, την κυβέρνηση τελικά, το, τοπικές αρχές, εθνικές αρχές, το, το, το έγκλημα και τα ναρκωτικά. Γι' αυτό και εγώ, εν κατακλείδη, θέλω να προτείνω σε γενικές γραμμές να υποστηρίξουμε τον κύριο Κόρτες για την εκθεσή του να κατεβάσουμε κάποιες τροπολογίες ούτως ώστε να βελτιωθεί το κείμενο τροπολογίες που θα έχουν την, το χαρακτήρα προσθήκης και όχι αντικατάστασης των διατάξεων του κειμένου. Επίσης, σε συνεργασία με τους άλλους Ισπανούς συναδέλφους, να δούμε πώς θα συνεχθούμε με το Υπουργείο Εξωτερικών, με ε, τις αντιπροσωπείες μας στο εξωτερικό και να μπορέσουμε επομένω έτσι να ασκήσουμε κάποια πίεση στο Συμβούλιο για να πάνε τα πράγματα προς την κατεύθυνση που σας εξήγησε ότι θέλουμε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στεμίρο. Πολύ θερητικά τα λόγια σας. Κύριος Γκέρινς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έφτασα καθυστερημένος και θα ήθελα απλώς να τοποθετηθώ στις, ε, στα σημεία 7 και 8 της, 8 της εκθέσεως ε, που μου φαίνονται από τα πιο λεπτά σημεία του θέματος αυτού. Εάν προσδιορίσουμε ως ε, κανόνα μας, ως αρχή μας την καταπολέμηση της φτώχειας, θα πρέπει να είμαστε και πλούσιοι για να βοηθήσουμε τους φτωχούς. Μην ξεχνάμε ότι τα χρήματα μπορεί να το... Και επίσης ότι ποιος θα διακρατά τα χρήματα. Μην ξεχνάμε ότι τα χρήματα μπορούν να τα διακρατούν τα κράτη χορηγία, αλλά μπορούν να τα διακρατούν και εκείνα τα οποία ήταν οι δικαιούχοι της ε, βοήθειας, αναπτυξιακής βοήθειας. Λοιπόν, τα δεδομένα τα, ε, της παγκοσμιοποίησης έχουν ανατρέψει τα πάντα. Οι διαφορές μέσα στα κράτη αλλάζουν ριζικά και πλέον η καταπολέμηση της φτώχειας είναι αρμοδιότητα της ίδιας της ε, κυβέρνησης. Εκείνη, εάν δεν τα καταφέρνει, πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες της γιατί δεν μπορεί να εξασφαλίζει την αναδιανομή του πλούτου έτσι ώστε να δώσει απαντήσεις στις θεμητές προσδοκίες των πολιτών. Δεν μπορούμε εμείς να υποκαταστήσουμε και να, την κυβέρνηση και να ε, αναλάβουμε 100% τις δικές τους ευθύνες. Αυτό πρέπει να το θέσουμε στην τράπεζα των συζητήσεων πλέον. Καλό την Επιτροπή να το πράξει. Εάν θέλουμε να δείχνουμε μια κάποια συνέπεια, είναι μια αρχή αυτή την οποία δεν μπορούμε να λησμονούμε. Πρέπει και να λαμβάνουμε υπόψη τι αλλαγέ και σε τελευταία ανάλυση το phasing out ε, είναι μια προοδευτική ε, μέθοδο, ένα μηχανισμό προοδευτικό, ο οποίο μα επιτρέπει να απεμπλακούμε διαδοχικά. Γι' αυτό λοιπόν καλό να σημειώσουμε ότι ναι μεν δεν πρόκειται να σταματήσει κάθε ε, συνεργασία από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά ε, πρέπει να αρχίσουμε και εμείς να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε σε 3, 5, 10 χρόνια από σήμερα. Διαφορετικά, σε τι εξυπηρετεί το midterm review, η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και όλη η δουλειά που κάναμε, στην οποία όλοι συμφωνήσαμε και αναγνωρίσαμε το ίδιο αυτό πρόβλημα που σας αναφέρω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντική παρατήρηση και χτες ακούστηκε η κάθε άστον χτες είπε ότι το triple down δεν φέρνει αποτελέσματα και άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε τα προβλήματα της, ε, των θυλάκων φτώχεια ε, σε χώρες όπου οι πλούσιοι καθίσανται όλο και πιο πλούσιοι ενώ οι φτωχοί είναι όλο και πιο φτωχοί και εσείς αμφισβητείτε το κατά πόσο είναι δική μας ευθύνη το να συμπληρώσουμε αυτό το κενό ή αν θα έπρεπε με τη δική μας ε, ε, επιρροή φυσικά και με την αξιοπιστία μπορούμε να προσφέρουμε στη διαδικασία αυτή να προχωρήσουν οι ίδιες οι κυβερνήσεις ε, και βέβαια μέσα από την εμπιστοσύνη σε διμερείς σχέσεις. Ο κύριος Γκόρισεκ τώρα παρακαλώ από το ΙΕΣ e θα ήθελα να αναφερθεί ειδικά στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και, Λατινοαμερ... και Λατινοαμερικανικών κρατών έτσι ώστε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις και ως προς τα όσα είπε ο κύριος και θα ήθελα επίσης να ακούσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Μπουλίτα Μπουτεβελίτσιεν και τον κύριο Ντελακαλάμπρια. Για το... Ζητώ συγγνώμη που σας σφαγίασα το όνομα. το μέσο DCI και τη συνεργασία λοιπόν επί τόπου. Ο κύριος Γκόρισεκ πρώτα όμως. Καλημέρα. και ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάστρα για την έκθεσή του, η οποία έρχεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή και καλύπτει όλα τα σημαντικά θέματα που περιλαμβάνει το προτινόμενο MFF και περιγράφει τη δομή της μελλοντικής μας συνεργασίας με την περιφέρεια. Έχουμε τα στοιχεία λοιπόν τα οποία θα μας επιτρέψουν να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Σε επίπεδο της διάρθρωσης, αυτό που διαφορο... η διαφοροποίηση είναι το πιο σημαντικό θέμα, όπως ανέφερε ένας από τους συναδέλφους σας ήδη. Αυτό που θα ήθελα να επαναλάβω είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση για μείωση της συνεργασίας με οποιαδήποτε από τις χώρες αυτές. Αυτό στο οποίο αναφερόμαστε είναι να μην χρησιμοποιήσουμε διμερεί κανάλια, αν θέλετε, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγχυση στην αντιμετώπιση και στην ανείχνευση των προβλημάτων στην ανάπτυξη. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν Έχουμε πολλά θέματα και μέσα, αν θέλετε, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο. Επί τη βάση λοιπόν των μαθημάτων που έχουμε πάρει από το παρελθόν, μπορούμε να φροντίσουμε τις χώρες της περιοχής, ακόμα και αυτές που έχουν σημαντικούς θύλακες φτώχειας. Και εδώ θα βασιστούμε, όπως είπε και ο κ. Ντεμέρα, σε κάποιες εμπειρίες τις οποίες ε, έχουμε συλλέξει από τις χώρες αυτές. Σε ένα σημείο της έκθεσης λέγεται ότι δεν θα πρέπει να μειώσουμε την βοήθεια προς τη Λατινική Αμερική. Αυτή είναι η πρόθεση της πρότασης. Δεν υπάρχει καμία σκέψη έτσι ώστε η μείωση, να υπάρξει μείωση σε σχέση με το παρελθόν. Για την ουσία τώρα της πρότασης ε, βλέπω με ικανοποίηση ότι τα περισσότερα στοιχεία της έκθεσης ε, α, μας βρίσκουν σύμφωνος. Έχουμε τρία θα έλεγα είδη στοιχείων. Πρώτον αυτά τα οποία μας βοηθούν να πετύχουμε τους κοινού στόχους, κοινωνική συνοχή και εκρίζωση της φτώχειας. Χρηστή διακυβέρνηση, φορολογικές πολιτικές, εκπαίδευση, υγεία, βοήθεια στις μικρομεσαίες, βοήθεια στις υποδομές και συνεργασία στην έρευνα και στην επιστήμη. Υπάρχουν επίσης και προβλήματα τα οποία βέβαια μας εμποδίζουν να πετύχουμε αυτούς τους στόχους που προανέφερα. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε στην εγκληματικότητα, στη βία που προέρχεται από το εμπόριο ε, ναρκωτικών. Είναι θέμα αυτό στην Νότια Αμερική και αν δεν το αντιμετωπίσουμε τότε δεν θα εκριζώσουμε πραγματικά τη φτώχεια. Απαιτούνται σωστές κοινωνικές πολιτικές, ενίσχυση της συνεργασίας, της δημοκρατίας, συγγνώμη, κλπ θέματα αυτά αν δεν τα φροντίσουμε θα έλεγα τότε οι στόχοι μας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν όπως επίσης και το θέμα της αντιμετώπισης των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Δύο επιπλέον θέματα. Πρώτον, διασφάλιση της συνεκτικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας και συμπερίληψη σε εισαγωγικά της κοινωνίας των πολιτών. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το DCI υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθούν τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης έτσι ώστε να διασφαλίσουμε και εμείς ως τότε χρήση των μέσων τα οποία διαθέτουμε. σε συγκεκριμένους τομείς μάλιστα για με στόχο τη σωστή συνεργασία με τις τοπικές πρωτοβουλίες και αρχές έχει υπάρξει και αύξηση των ε, πιστώσεων. Προσπαθήσαμε στα πλαίσια του ισχύοντος DCI να προωθήσουμε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Μερικές φορές αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και λόγω των δικών μας πρακτικών συνειδητοποίησαμε λοιπόν ποιες είναι οι δυσκολίες αυτές και χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτή τη μορφή συνεργασίας και εκμεταλλευόμενοι τις θετικές εμπειρίες σε ορισμένες χώρες προσπαθήσαμε να τις μεταφέρουμε σε άλλες χώρες της περιοχής βελτιώνοντας γενικά την συνεργασία στα πλαίσια πάντα των γενικών αρχών. Ευχαριστώ κύριε Γκόρισεκ. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπετε ότι είμαι για πρώτη φορά εδώ. Σημείωσα ότι ακούστηκε μέχρι τώρα. Κύριε Κορτές Λάστρα, χαίρομαι που σας συναντώ ε, διάβασα την εκθεσή σας, μου προκάλεσε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, όλοι οι φίλοι της Λατινικής Αμερικής ε, πρέπει να βοηθήσουν. Εμείς εκτιμήσαμε το περιεχόμενο των προτάσεών σας και την πρόσκλησή σας για το πώς μπορούν όλα αυτά να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα. Δεν θα διαφωνήσω με αυτά που ακούστηκαν, είναι πάρα πολύ λογικά. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα όταν προσπαθεί κανείς να εφαρμόσει τις πολιτικές αυτές επί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα ήταν αξιόπιστη αν χρησιμοποιούσε πάντα τους ίδιους τρόπους και τις ίδιες μεθόδους. Πράγματι για πάρα πολλά χρόνια με πολλούς εταίρους κάνουμε τα ίδια πράγματα αλλά πολλές φορές κάνοντας το αυτό δεν φτάνουμε στους βαθύτατους θύλακες φτώχειας. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να επανατοποθετηθούμε Ξέρετε ότι υπάρχει πλέον μια οικονομική πίεση θα έλεγα, προσπαθούμε να είμαστε ειλικρινεί, προσπαθούμε να βρούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς να πείσουμε τους εταίρους μας έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις μορφές παρέμβασής μας. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι στα ειδικά χαρακτηριστικά της Νοτιού Αμερικής. Προφανώς τα θέματα ασφαλείας ή ανασφάλειας που υπάρχουν εκεί δεν υπάρχουν σε άλλες περιοχές να αναφερθώ πάρα πολύ σύντομα σε αυτά τα οποία ανέφερε η κυρία Κέλλερ. Όταν αναφερόμαστε στα θέματα ασφαλείας, αναφερθήκατε στην ατιμορρησία, στα θέματα της δικαιοσύνης. Συνδέεται λοιπόν το θέμα της δικαιοσύνης με την ασφάλεια. Το θέμα της αποκατάστασης του συστήματος, ε, ε, ε, αποκατάστασης του δικαστικού συστήματος δεν είναι κάτι το οποίο σώνει και καλά οδηγεί αποκλειστικά στη χρηματοδότηση νέων σοφρονιστικών καταστημάτων. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος. Προσπαθούμε να παρέμβουμε σε τομείς όπως η εκπαίδευση στο Σελ Σαλβαντόρ. Οι γονείς είναι ελεύθεροι να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία Δυστυχώς όμως το ποσοστό εγκατάλειψης είναι πάρα πολύ υψηλό. Έχουν τα μέσα, έχουν τα βιβλία, έχουν τους δασκάλους, αλλά φοβούνται οι γονείς μερικές φορές να στέλνουν τα παιδιά για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να γνωρίζουμε την πραγματικότητα, πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς πρωταγωνιστές και να εξυπηρετούμε έτσι και τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Προσπαθούμε να βρούμε και νέους τρόπους για να ενταχθούμε στον λεγόμενο χώρο της ανάπτυξης. Το νέο μέσο που λέγεται μέσο για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στη Λατινική Αμερική. Οι ανάγκες οι επενδυτικές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Με δάνεια μόνο δεν μπορεί κανείς να πετύχει τους στόχους. Προσπαθούμε πώς μπορούμε να αναμίξουμε εμείς δάνεια, πιστώσεις, με ιδιωτικές επενδύσεις και αναπτυξιακά δάνεια έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους της ανάπτυξης. Κάποτε ας πούμε αγαπούσαμε να φτιάχνουμε δρόμους. Ε, γιατί τώρα να φτιάχνουμε βέβαια κάποιους δρόμους στην Ποτσουάνα οι οποίοι δεν πηγαίνουν πουθενά. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι ο δωρητής ε, ε, χαίρεται όταν βλέπει να πιάνουν τόπο τα χρήματα τα οποία δίνει. Λοιπόν, υπάρχουν εδώ ανάγκες για ενημέρωση δεν υπάρχουν ε, πάρα πολλές δυνατότητες για δημιουργία δρόμων πλέον μέσω των δικών μας μορφών χρηματοδοτήσεων. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε υποδομές οι οποίες είναι άχρηστες. Παρόλα αυτά πρέπει να βοηθάμε να αναπτύσσονται οι δευτερογενείς οδικές συνδέσεις που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της υπαίθρου. Σαν παράδειγμα, ε, οικοδομούμε ανεμόμυλους στο Μεξικό. Πού το κάνουμε αυτό, το κάνουμε σε περιοχές όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι τοπικοί ηθαγενείς πληθυσμοί. Ε, δεν είναι εύκολο να προχωρούμε σε αυτές τις ε, ενέργειες. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τις τοπικές ανάγκες με τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Σαν παράδειγμα, για το συγκεκριμένο πλαίσιο έχουμε 125 εκατομμύρια διαθέσιμα και προκάλεσαν 5 δις ε, επενδύσεις. Έχουμε λοιπόν εδώ απόδοση της προσπάθειάς μας και μπορούμε να βοηθήσουμε και προγράμματα στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα του περιβάλλοντος κτλ. Αν μακρηγορώ να μου πείτε να σταματήσω. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Γκέρεντς για την παρέμβασή του. Υποστηρίζει την άποψη που εκφράσαμε ότι πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι αλλάζοντας κάποια από τις μεθόδους μας. Δεν θα πρέπει να αλλάζουμε συνεχώς βέβαια, αλλά θα πρέπει να αλλάζουμε και να προσαρμόζουμε τις μεθόδους μας. Η πιο αγαπημένη μου χώρα, η Κολομβία, περίπλοκη χώρα, Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα αυτή, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τον Ερυθρό Σταυρό. Είναι προφανές θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την κοινωνία των πολιτών. Αυτό δεν χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα βέβαια. Ίσως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διμερεί προγράμματα με διαφορετικό τρόπο και έτσι να βοηθήσουμε και τις υπόλοιπες χώρες ε, της κοινότητας των Άνδεων Ίσως τα λέω λίγο τεχνικά, αλλά συμφωνώ με την άποψή σας ε, ότι πρέπει να ενισχύσουμε την παρέμβασή μας στην περιοχή. Όταν συνάντησε τον πρόεδρο Σάντος ο Επίτροπος Πίμπαλτς είπε ότι εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε ε, ας προσπαθήσετε να μείνετε ε, στο πλάι μας για κάποιες μικρές ακόμα χρονικές περιόδους και τα πράγματα ε, θα βελτιωθούν και θα αυξηθούν και οι διαθέσιμες πιστώσεις και στον τομέα της δικαιοσύνης και στον τομέα της αντιμετώπισης του φαινομένου της ατιμορρησίας θα υπάρξουν πιστώσεις για όλες τις χώρες της Συμφωνίας των Άνδεων. Δεν αλλάζουμε συνεχώς άποψη, Αντιμετωπίζουμε όμως νέες μεθόδους, την πιθανότητα εφαρμογής νέων μεθόδων. Αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα το συζητήσετε στα πλαίσια του MFF για το DCI, οι ανάγκες συνεχίζουν να υπάρχουν και δεν μειούνται οι, ε, οι ανάγκες αυτές. Εντυπωσιάζει να βλέπει κανείς ότι οι πιο, δίκαιες χώρες, η πιο δίκαια χώρα θα έλεγα ε, στη Νότια Αμερική είναι η Ουρουγουάη, παρόλα αυτά έχει τρομερές κοινωνικές ε, εσωτερικές διαφορές. Λοιπόν, ε, υπάρχουν πολλά τα οποία μένει να γίνουν, συνεργαζόμαστε με τις χώρες αυτές σε υψηλό επίπεδο, με υπουργούς από τις αναπτυσσόμενες χώρες, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και αυτόν τον τομέα. Συνειδητοποιούμε λοιπόν τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, εκτιμούμε τις προτάσεις οι οποίες ακούστηκαν μέχρι τώρα, σημείωσα τις προτάσεις τις οποίες κάνατε και να είστε βέβαιοι ότι θα προσπαθήσουμε να τις ε, κάνουμε πραγματικότητα. Συναντηθήκαμε με τους ομολόγους μας στην Ισπανία και με την Γερμανία στον τομέα της ανάπτυξης και συζητήσαμε μαζί τους για το πώς μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε τη δική μας παρέμβαση, πώς μπορούμε να φέρουμε στη συζήτηση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μην αγνοήσουμε τα κοινωνικά θέματα, να μην αγνοήσουμε το θέμα της υγείας, όταν θα υπάρξει αυτό το, αυτή η νέα στην αντιμετώπιση των θεμάτων της Λατινικής Αμερικής. Ευχαριστώ πολύ. Η καλύτερη παρουσίαση από την Επιτροπή το τελευταίο καιρό. Πολύ συγκεκριμένη για τα προγράμματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλος από την Επιτροπή. Ρικάρντο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους και ιδιαίτερος για την υποστήριξη στην ε, δουλειά αυτή, στην έκθεση. Σε έναν βαθμό τουλάχιστον θα ήθελα να πω ότι αυτή η έκθεση αποτελεί καρπό όλων των εργασιών που έχουμε κάνει εδώ, των συνεδριάσεων, ε, με την ΕΝΤΕΦΚΟ, με τα Ηνωμένα Έθνη, την Κοινωνία των Πολιτών, την Υπηρεσία Εξωτερική Δράσεω. Αποτελεί ένα πρώτο σκαρίφημα των όσων έχουμε πει. Και τον κύριο Φίσα, τον οποίο θα ήθελα θερμά να ευχαριστώ γιατί έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά και έχει συμβάλει πολύ στην έκθεση αυτή. Είναι μια έκθεση λοιπόν κοινή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους ε, για την ε, ιδιαίτερη ευαισθησία που δείχνουν για τη Λατινική Αμερική και την βαθιά γνώση του θέματος. Σε μια περίοδο τόσο σημαντική και στρατηγική σημασία αυτή τη στιγμή ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε πάνω απ' όλα την ε, ορατότητα για μια σταδιακή μείωση του DCI, όχι δηλαδή απότομη διακοπή, για να εξηγήσουμε και να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα το θέμα αυτό. Και θέλω να πω στον κύριο Γκέρνσο στο σημείο 10 της εκθέσεως, όπως γνωρίζετε, μιλάμε για συγχρηματοδότηση προγραμμάτων δεν χρηματοδοτούμε, αλλά συγχρηματοδοτούμε. Ευχαριστώ την κυρία Κέλλερ. Και συμμερίζομαι σωστικά όλα τις τα σχόλια. Θα συνεργαστούμε και με τον κύριο Σαντιάγο Φίσας, όπως και με την κυρία Κέλλερ, ε, για τις τροπολογίες. Για τον κύριο Γκέρενς ήθελα απλώς να υπογραμμίσω την συγχρηματοδότηση για την σημαντική. Και Μερικά σχόλια, αν μου επιτρέπετε, προς την Επιτροπή σε σχέση με τα δύο θέματα που γνωρίζουμε, πιστεύουμε κάπως, την ασφάλεια καταρχάς και το λαθρομπόρο των ναρκωτικών, γιατί έχουμε συζητήσει μέσα από ένα σεμινάριο υψηλού επέδου στο Μεξικό τυχαία. Δεν ήταν εσκεμμένη η επιλογή. Ε, συζητήσαμε το θέμα του ε, ναρκωτικών και βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο δράσης που δεν αντιστοιχεί ενδεχομένω στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τη Επιτροπή μα, αλλά πάντως μας εντυπωσίασε η κατάσταση όχι μόνο στη Λατινική Αμερική, αλλά εν γέννη ε, με πολλές χώρες δυνατότητα για συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών, για ανάπτυξη ουσιαστική δουλειά δουλειάς καταπολέμησης της ε, ε, καταπολέμησης της, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Απέχουμε έτη φωτός από τη δικαστική συνδρομή που χρειάζεται για να μπορέσουμε να κάνουμε μια πραγματική ε, να, έχουμε ένα πραγματικό αποτέλεσμα στην πάταξη του λαθρεμπορίου ναρκωτικών από, σε συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής. Άλλωστε εδώ επαναρχόμαστε στο πρόβλημα της κυρίας που επισήμανε και η κυρία Κέλλερ. Νομίζω ότι εμείς έχουμε να προσφέρουμε ένα σημαντικό know-how ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση θα έλεγα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε, το λέω και στην Υπηρεσία Ευρωπαϊκή ε, Εξωτερική Δράση και στην ΕΔΕΦΚΟ, ότι πρέπει να παραμείνει αυτή η θέση, πρέπει να εμείνουμε και το phasing out, η διαδικασία αυτή είναι μια λογική διαδικασία. Έχουμε εντατική συνεργασία τα τελευταία χρόνια με τα κράτη αυτά. Έχουμε συνεργαστεί μέσα σε συμφωνίε σύνδεση, έχουμε συζητήσει ουσιαστικά και έχουμε, αποτύχει, έχουμε επιτύχει αποτελέσματα. Δεν μπορούν ξαφνικά κάποια κράτη από αυτά, με δείκτες μάλιστα ορισμένα εξ αυτών ε, πολύ εντυπωσιακού. Κολομβία, Εκουαδόρ, Περού ειδικά να μας φέρουν προ ε, τέτοιων εκπλήξεων με την απόφαση που έλαβαν, η οποία είναι πιστεύω και πρόημη και μπορεί να επηρεάσει ουσιαστική δουλειά που έχει γίνει εδώ και μήνες και που έχει να κάνει ιδιαίτερα με τις αδυναμίες που εντοπίζονται στην περιοχή αυτή. Το ότι ορισμένες χώρες τώρα λένε ότι έχουν μακροοικονομική συνθήκη και ανάπτυξη μακροοικονομική σημαίνει ότι γνωρίζουν ποια είναι τα προβλήματά του. Θα έπρεπε να γνωρίζουν όμως τα προβλήματα και στον τομέα της δικαιοσύνης, ε, της κοινωνικής συνοχής, της εκπαίδευσης, της ε, δημόσιας υγείας. Εμείς με την τεχνογνωσία και το δυναμικό που έχουμε ε, να προσφέρουμε, αποδεικνύουμε ότι οι πόροι που έχουμε προσφέρει στην αναπτυξιακή συνεργασία φέρνουν καρπούς, έχουν φέρει καρπούς και έχουν στηρίξει μια περιοχή με την οποία έχουμε συνεργαστεί σε ουσιαστικά, ε, στην, επιτυχάνοντας ουσιαστικά αποτελέσματα. Ακόμη και ως χορηγή αναπτυξιακής βοήθειας μπορούμε να συνεργαστούμε με τα κράτη αυτά μέσα σε μια τριγωνική σχέση που θα μπορέσει να αποτελέσει το μέλλον της αναπτυξιακής συνεργασίας στην Ευρώπη. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η σταδιακή μείωση τετραετής. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε για μερικά χρόνια ακόμη και όπως υπόθηκε και νωρίτερα να δείξουμε ότι υπάρχει μια προοπτική και παραμένουμε ε, στην περιοχή αυτή ε, ακόμα παρόντες. Πολλά ακόμα μπορούμε να κάνουμε στη συνεργασία μας με τα κράτη αυτά και ιδιαίτερα όταν έχουμε μια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε μια μέρα στην άλλη την περιοχή αυτή, τη Λατινική Αμερική δηλαδή. Ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία σα για όλε τι καλέ ιδέε. Και περιμένω να δω και νέε προτάσει για καλή συνεργασία, ώστε να βελτιώσουμε την έκθεση κατά τρόπον ώστε να ικανοποιεί στο μέγιστο δυνατό τι προστερές ομάδες τη ε, επιτροπή μα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κορτές Λάστρα. Και πριν ε, κλείσουμε, θα ήθελα να πω από τα όσα είδαμε σήμερα στη συζήτησή μας, από τα όσα μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι όλα αυτά που ανακοινώθηκαν θα πρέπει να ε, συνδεθούν στενά με τις διαπραγματεύσεις της ΣΥΑΕ που θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με το Συμβούλιο μια ιδιαίτερη δηλαδή ομάδα ανθρώπων που θα έχουν την ευθύνη αυτών των διαπραγματεύσεων, ειδικοί, με τους οποίους θα πρέπει να συνεργαστείτε εσείς, ώστε να βεβαιώνεστε κάθε φορά ότι και οι προτεραιότητες που έχετε προσδορίσει στην έκθεση σας λαμβάνονται υπόψη κατά τι συζητήσει και διαβουλεύσει για την εφαρμογή του DCI με το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Οι τροπολογίες προβλέπεται να κατατίθεται μέχρι τις 19 Μαρτίου, ψηφοφορία στις 24 και θα ήθελα τεχνικά για ένα τεχνικό ζήτημα να επισημάνω ότι το ICD πρέπει να λέγεται DCI. Αυτό που στο αγγλικό κείμενο λέγεται ICD θα πρέπει να το διαβάζουμε DCI, θα γίνει σχετική τροποποίηση στην Ολομέλεια. Και το επόμενο μας θέμα είναι ο ρόλος των κοινοβουλίων στο να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του προγράμματος δράσης υπέρ των λιγότερων επιτυγμένων χωρών για τη δεκαετία 2011-2020. Έχουμε τη Διακοινοβουλευτική Ένωση και τους εκπροσώπους της. Η κυρία Νόρα Μπάμπεκ ε, από την Διακοινοβουλευτική Ένωση έχει έρθει εδώ για να συστήσουμε την τέταρτη έκθεση για τη δεύτερη, τέταρτη διάσκεψη των Αθηνών για τις λιγότερες, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, μια διάσκεψη που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη πέρυσι. Η κυρία Μπάμπικ ε, είναι ε, μεταξύ των ε, αρμοδίων για το πρόγραμμα IPU, Institutional Capacity Building δηλαδή, και ασχολείται ιδιαίτερα με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τη δυνατότητα για έλεγχο και λογοδοσία των κυβερνήσεων των χωρών αυτών ως προς τη δαπάνη, την χρήση των κονδυλίων. Αυτό μέσα σε μια ενισχυμένη συνεργασία απευθύνεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες, στις LCD δηλαδή, χώρες ε, με τα περισσότερα προβλήματα, 48 τον αριθμό, αυτές που έχουν χαμηλό ε, κατακεφαλήν εισόδημα καθυστέρηση ανάπτυξη και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα ευάλωτε ε, στις ε, διάφορους, κλειδονισμού στην εσωτερική αλλά και εξωτερική αστάθεια και χρειάζονται το, το, πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ώστε να αναπτύξουν την οικονομική του ανάπτυξη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα δράση, το πρόγραμμα δράση των Βρυξελών, ένα νέο πρόγραμμα δράση. Τώρα προσδιορίζει νέα προσκόμματα, νέε προκλήσει και δυνατότητε για τι λιγότερο επιτυχημένε χώρε και του χορηγού. Πέραν αυτών ε, υπάρχουν και τρεις παράλληλες ε, δομές κυβερνητική κοινωνία των πολιτών και ιδιωτικό τομέα, παράλληλη με τη διάσκεψη τη Κωνσταντινούπολη. Αυτή η τρίτη διάσκεψη για τι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε των Βρυξελών του 2001 είχε, είχε επίσης αποτελέσει μια ε, ευκαιρία για νέες και επικοδομητικές συνεργασίες με το πρόγραμμα δράσης των Βρυξελών, ιδιαίτερα στον χώρο της ε, ορθής διακυβέρνησης και της ανάπτυξης δυναμικού και έχει, αναπτύξει, έχει ανοίξει το δρόμο για την διάσκεψη Κωνσταντινούπολης. Εγώ ήμουν παρόν εκεί. Ήταν πολύ εντυπωσιακή η συνεδρίαση. Αποτέλεσε σημαντική ε, συμβολή στην ε, εμπλοκή στον αγώνα για την ε, καταπολέμηση των προβλημάτων των λιγότερων ανεπτυγμένων κρατών, follow-up εφαρμογή του νέου προγράμματος δράσεως για τις χώρες αυτές μετά το 2011 και το 2020. Βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί πλήρως την εφαρμογή και την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος δράσεως Κωνσταντινούπολης και αν μου επιτρέπετε τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπαμπίκ. Ευχαριστώ αγαπητά μέλη. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας σήμερα αντιπροσωπεύοντας τη Διακοινοβουλευτική Ένωση και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για την κοινοβουλευτική συνεισφορά στο πρόγραμμα της Κωνσταντινούπολης η κοινοβουλευτική πλευρά αν θέλετε ξεκίνησε να αναπτύσσεται εδώ και τέσσερα χρόνια θα πρέπει και για τις διασκέψεις για τις λιγότερο προχωρημένες χώρες, αναπτυγμένες χώρες, να ακουστούν και οι απόψεις των κοινοβουλευτικών. Τα τελευταία χρόνια τα κοινοβούλια θεωρούνται θεωρητικά για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των Βρυξελών. Αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα έχει αλλάξει. Το πρόγραμμα δράσης αναφέρεται στο ρόλο των κοινοβουλίων και στην ανάπτυξη προγραμμάτων για τις υποανάπτυξη χώρες στηρίζοντας την συμμετοχή και τη διαφάνεια. Χάρη ακριβώς στους βουλευτές οι οποίοι έκαναν προσπάθειες για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν νέες προοπτικές για τις υποανάπτυξη χώρες. Πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά α, τους λαούς των χωρών ανεξαρτήτως του κοινωνικού καθεστώτος, ανεξαρτήτως του φύλου, επιτρέποντας να πάρουν μέρος στην προσπάθεια. Το πρόβλημα της ανάπτυξης είναι πολιτικό και όχι οικονομικό. Υπό ανάπτυξη χώρες είναι 880 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν τεράστιες δυνατότητες στον πολιτισμό και σε φυσικούς πόρους. Το θέμα είναι ποιος αποφασίζει και για ποιον ποιος ε, παίρνει τις αποφάσεις και στο όνομα ποιου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε επίπεδο κοινοβουλίων και σε επίπεδο κυβερνήσεων και σε επίπεδο διεθνών οικονομικών οργανισμών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ίσως όμως να υπάρχουν και κάποιες άλλες δυνατότητες. Θέλουμε να ξεκινήσουν με μια νέα όφηση οι οικονομίες αυτές τις χώρες. Ας πάρουν και οι γυναίκες τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι άνδρες για να αγοράζουν γη ή να παίρνουν δάνεια. Θέλουμε οι φτωχοί να ξεφύγουν από τον ανεπίσημο τομέα και να περάσουν σε μικρές επιχειρήσεις και σε θέσεις με σωστούς μισθούς. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να τους βοηθήσουμε να παίρνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ή να δημιουργούν συνδικάτα. Θέλουμε οι χώρες να βοηθηθούν από τους φυσικούς τους πόρους. Ε, θα πρέπει οι φυσικοί πόροι να μην γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω διεφθαρμένων θα έλεγα συστημάτων και ε, να ωφελούνται μόνο ε, ομάδες συμφερόντων στο εξωτερικό. Ας ενισχύσουμε και τα πολιτικά μας μέσα. Αυτό σημαίνει ότι τα πολιτικά κόμματα και τα, ελεκτι τα συστήματα τα εκλογικά πρέπει να βελτιωθούν χωρίς να υπάρχει χρήση βίας. Θέλουμε η ξένη βοήθεια να χρησιμοποιείται με τον καλύτερο τρόπο σύμφωνα με τις προτεραιότητες. Ας είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι η βοήθεια ελέγχεται κοινοβουλευτικά και σε επίπεδο δωρητριών χωρών και σε επίπεδο αποδεκτών. Ε, το θέμα δεν είναι να αρνηθούμε την οικονομική πραγματικότητα, αλλά τα οικονομικά προβλήματα συνδέονται με μεγάλα θέματα αντιπροσώπευσης, συμπερίληψης και επίσης του να είναι κανείς υπόλογος. Η κυβέρνηση πρέπει να είναι η υπόλογη ακόμα και στην ομοθετική της δραστηριότητα και όχι μόνο στην εφαρμογή των νόμων. Η διακυβέρνηση είναι θα έλεγα στην καρδιά του κοινοβουλευτικού μηνύματος το οποίο υπέβαλαν τα μέλη της IPU στην διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης. Ανάμεσα σε άλλα το έγγραφο της IPU ζητάει από όλα τα κοινοβούλια και από τις χώρες LDC και από τις χώρες μη LDC να ελέγξουν τις θεσμικές διαδικασίες τις οποίες ακολουθούν σε σχέση με τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Απαιτούνται στενότερες σχέσεις βέβαια ανάμεσα στους εμπλεκομένους. Αυτό θα εξαρτηθεί και από τις δυνατότητες που έχουν οι ίδιες οι χώρες έλντιση ε, και έτσι θα πιέσουν και την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Τώρα είμαστε στα πλαίσια της συζήτησης σαν κοινοβούλια θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την εφαρμογή. Το IPA δεν είναι τέλειο και δεν περιλαμβάνει αρκετούς στόχους, αλλά είναι ένας ξεκάθαρος δρόμος για τα επόμενα δέκα χρόνια. Βασικός μας στόχος είναι να γίνει mainstreaming του IPOA μέσω εθνικών αναπτυξιακών στρατηγικών εδώ και 10 χρόνια, 10 χρόνια μάλλον θα περάσουν γρήγορα και ήδη πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε το μέλλον στον τομέα των κοινοβουλίων. Στα πλαίσια πάντα του IPOA, σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Εξωτερικών, ε, εξωτερικών Σχέσεων. Βασικός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε τις προσπάθειες που κάνουν τα κοινοβούλια γνωρίζοντας ποια είναι τα στοιχεία τα οποία προτείνει το IPOA. Αυτό ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο. Σε πάρα πολλά κοινοβούλια, ιδιαίτερα στις χώρες LDC, δεν υπάρχουν ενημερώσεις σωστές των κυβερνήσεων ή από πλευρά των κυβερνήσεων για τις διεθνείς συμφωνίες, τις αναπτυξιακές τα μακροπρόθεσμα θα έλεγα, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του συστήματος είναι να διασφαλίσουμε την εμπλοκή των κοινοβουλίων, να ενημερώσουμε σωστά τα κοινοβούλια και να ενισχύσουμε τις δυνατότητες που έχουν τα κοινοβούλια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Βράχει πρόθεσμα θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες μεθόδους επικοινωνίας ανάμεσα στις χώρες LDC και στις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιώντας τους εξειδικευμένους μηχανισμούς που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμοι. Προσπαθούμε επίσης και να καλύψουμε τις ανάγκες ορισμένων κομβικών θεμάτων για τα οποία ειδικά τα κοινοβούλια πρέπει να δώσουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο τομέας σαν παράδειγμα των θεσμικών τρόπων λειτουργίας, έτσι ώστε να εντάσσονται τα κοινοβούλια στις πολιτικές, νομοθετικές και δημοσιονομικές διαδικασίες. Θέλουμε τα κοινοβούλια των χωρών αυτών να υιοθετήσουν ένα πρόγραμμα δράσης έτσι ώστε να εξηγήσουν σαφώς τον τρόπο απορρόφησης του IPOA Πολλά κοινοβούλια πήραν μέρος τον προηγούμενο Μάιο στη διακοινοβουλευτική συνάντηση της Κωνσταντινούπολης και είναι ήδη ενήμερα. Υπάρχει ένας κατάλογος των βασικών προγραμματικών θα έλεγα δραστηριοτήτων. Δεν θα επιμείνω, αν θέλετε επιπλέον πληροφορίες να σας τις δώσω. Πέρα από τις δραστηριότητες αυτές όμως Προσπαθούμε να ενισχύσουμε και την, βοήθ την προσπάθεια συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων που έχουν τα κοινοβούλια. Τον προηγούμενο Οκτώβριο είχαμε την βασική ενημέρωση των βουλευτών μετά από τη διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης έτσι ώστε κάποια από τα μηνύματα εν περιπτώσει ε, που περιλαμβάνει το IPOA να γίνουν κατανοητά. και στον τομέα του mainstreaming. Είπαμε τα υπέρ και τα κατά της δημιουργίας νέων κοινοβουλευτικών δομών που θα εξετάσουν τις προτάσεις αυτές παράλληλα με τις υπάρχουσες δομές. Λοιπόν, για την αηφορία τώρα και πού βρίσκεται η αηφορία για τα κοινοβούλια αυτά των χωρών LDC. Ελπίζουμε τα κοινοβούλια να αποκτήσουν τους κατάλληλους μηχανισμούς, να ενημερώνονται σωστά και να συνεργάζονται με τις εθνικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τα προβλήματα της ανάπτυξης. πρέπει να προωθηθεί στα πλαίσια του IPU η περαιτέρω επικοινωνία ανάμεσα στα κοινοβούλια. Έχουμε 35 κοινοβούλια που είναι μέλη της IPU σήμερα από πλευράς των χωρών αυτών και συναντώμεθα μαζί τους τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Θα ζητήσουμε τη στήριξη του προγράμματος και σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και Κοινωνίας των Πολιτών. Η στρατηγική της εταιρικής σχέσης μας οδηγεί στη συνεργασία με τον είπα το εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο προχωρημένες χώρες οικονομικά και ελπίζουμε έτσι να εφαρμόσουμε σωστά το πρόγραμμα δράσης υπογραμμίζοντας τον ρόλο των κοινοβουλίων που δεν ήταν ξεκάθαρο στο παρελθόν. Τα κοινοβούλια και στις χώρες LDC και στις χώρες ε, μη που δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτή πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε επίπεδο περιφερειακό και υποπεριφερειακό. Υπάρχει ένα σύστημα κόμβων το οποίο έχει ε, διευκρινιστεί και σε επίπεδο υπουργικό και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Εμείς στο IPU, στην ε, Διακοινοβουλευτική Ένωση, έχουμε δημιουργήσει τα φόρα μέσα στα οποία όλες οι πλευρές θα συζητούν την εφαρμογή του προγράμματος της Κωνσταντινούπολης και θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες και στον τομέα της επικοινωνίας με την κοινωνία των πολιτών Προσέθεσα εδώ κάτι που είπε ένας από τους ιδρυτές της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Ένωσης που έχει άμεση σχέση με τις χώρες αυτές και τα κοινοβουλιά τους. Ο κόσμος σήμερα είναι φτιαγμένος από πραγματομένες θα έλεγε κανείς ουτοπίες. Η σημερινή ουτοπία είναι η αυριανή πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να τολμήσουμε και στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Ο κύριος Ντίβα λέγει ότι σας ευχαριστώ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Δεν ξέρω αν κυρία Μπάμπιτς ξέρετε ότι και στο δικό μας κοινοβούλιο έχουμε μία υπηρεσία για την πρόθεση του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος από την υπηρεσία αυτή παρόν εδώ σήμερα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι παρόντες, θα έπρεπε να είναι. Και θα πρέπει να έρθετε σε επαφή και με, το, με την δική μας αυτή υπηρεσία, ίσως και ήδη να το κάνετε. Δεν ξέρω όχι για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, αλλά με το PPD του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανταλλάσσουμε θέματα για άλλα θέματα. Θα το θέσω το θέμα και αυτό στις επαφές ε, ε, μαζί τους. Ο κύριος Κάτσμαρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε. Βεβαίως και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορέσουν να συμμετάσχουν βουλευτές από τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Στις ε, ισομερείς κοινοβουλευτικές ε, συνελεύσεις έχουμε διαπιστώσει το πόσο χρήσιμες είναι τέτοιες συναντήσεις. Αυτή η διακοινοβουλευτική ένωση διόρμεται σημαντικό ρόλο στη ΔΕΠΟΛΟΝΙΑ ο βασικός τρόπος επαφής είναι διμερείς ομάδες επαφής, τις λέμε. Και κάθισα και ρώτησα τους ε, Πολωνούς συναδέλφους αν ε, είναι ενημερωμένοι για όλα αυτά Οι περισσότεροι δεν ήταν. Δεν ξέραν για αυτούς τους φορείς, για αυτά τα σχήματα. Και τελικά μόλις ένα 4% ε, ξέρει, ασχολείται με τα ζητήματα αυτά. Τα αναπτυξιακά αυτά ζητήματα και για τους στόχους της χιλιετίας και επομένως θα πρέπει να αυξηθεί και η προς αυτές τις ε, δραστηριότητες και άρα θα πρέπει να ενημερώσουμε τους ε, βουλευτές για όλα αυτά και σε βελτιωθεί και η κατάσταση επί την πολιτική αυτή. Κυρία Κέλλερ, έχετε το λόγο λέει ο πρόεδρος. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και για την ε, εισήγηση. Να δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά την εφαρμογή αυτού αυτής της διακήρυξης, της δήλωσης της Κωνσταντινόπολης. Βεβαίω και υπάρχουν και κάποια όρια σε σχέση με το πόσα χρήματα μπορούμε να δαπανίσουμε για τέτοια μέσα πολιτική Πάντως, μπορούμε να κάνουμε κάποια ουσιαστικά πράγματα και πρώτα-πρώτα να διαπιστώσουμε ότι μπορούμε να επηρεάσουμε και με την Επιτροπή και την ε, Πολιτική Γεωργίας και με την ε, Πολιτική Αλίας έτσι μπορούμε να πετύχουμε τις προτεραιότητες μας για τους ε, στόχους και της Κωνσταντινούπολης και τους αναπτυξιακούς θα πρέπει όμως να απευθυνθούμε και στις άλλες κοινοβουλευτικές επιτρόπες Δεν είναι εύκολο το έργο μας αυτό το εμπιστώσαμε και στο παρελθόν. Όμως θα πρέπει όλα αυτά να αποτελέσουν υψηλές προτεραιότητες. Γιατί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Δεύτερον. Βεβαίω και οι κυβερνήσει του, όλοι, όλοι θα πρέπει να συμβάλλουν στην υλοποίηση. Όλοι θα πρέπει να τηρήσουν τι υποσχέσει του. έχουμε δεδομένες τις δεσμεύσεις μας για την αποτελεσματικότητα της εμπειρεξιακής βοήθειας, επομένως να τηρηθούν από όλους τα υπεσχημένα. Εντάξει, ούτε ε, τα ξέρουμε όλα, ούτε μπορούμε να είμαστε παντού. Και παράλληλα έχουμε και την τακτική ε, κοινωνική μας εργασία. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Θέλει άλλο το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα, ευχαριστώ για την τόσο ενδιαφέρουσα εισήγηση από την εκπρόσωπο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. Βεβαίω και θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση στα κοινοβούλια για την ε, δήλωση της ε, Κωνσταντινούπολης και την ε, ανάγκη εφαρμογής της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί και αυτή να βοηθήσει και είναι αποφασισμένη να υποστηρίξει τις λιγότερο εμπληγμένες χώρες και ούτως ώστε οι φιλόδοξοι στόχοι της Κωνσταντινούπολης να επιτευχθούν. Επίσης, θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια που έχουμε για την πολιτική μέχρι το 2020 για αυτές τις χώρες. Είναι επίσης σημαντικό όμως το να πάρουν και τις στιγμές τους στα χέρια τους την πρωτοβουλία αυτές οι χώρες. Εμείς θα είμαστε ένας δυναμικός εταίρος τους. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε μια σωστή εφαρμογή του οράματος της Κωνσταντινούπολης με τα κατάλληλα προγράμματα. Εμείς θα σας ενημερώνουμε όσο γίνεται πληρέστερα. Ευχαριστώ. I'm Θα δώσω τον λόγο του ο Πρόεδρος στον κύριο Μίτσελ γιατί να μας μιλήσει. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστούμε και για την εισήγηση. Ίσως δεν το θεωρείτε τόσο σημαντικό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Τώρα έχουμε σε επαφή με τους βουλευτές από εκείνες τις ε, χώρες. Όποτε λοιπόν τους συναντούμε. Διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές δεν έχουν τη στοιχειώδη ενημέρωση. Ούτε έχουν τα κατάλληλα μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους. Συνήθηκα με έναν συνάδελφο από κάποια αφρικανική χώρα και δεν είχε ούτε καν συνεργάτη να τον βοηθάει. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με, το τα με τις αποστολές, ποια είναι τα προβλήματα. Πολλές φορές πάμε σε, σε μέρη τα οποία δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. πολλές φορές μόνο εκεί πέρα υπάρχει μεγάλη φτώχεια και επομένως ε, ενδιαφέρομαι μεν να πάω κάπου για να βοηθήσω αλλά να, να βοηθάω γι' αυτό και δεν έχω χρησιμοποιήσει καν τα χρήματα τα οποία μας διατίθενται για ταξίδι Άρα Ας είμαστε πιο δραστήριοι στην ενημέρωση για το πόσο σημαντική είναι αυτή η αναπτυξιακή πολιτική. Πρόεδρος, σε ευχαριστώ, έχεις δίκιο. Στο Κοινοβούλιο ε, προσπαθούμε, δική μου υπηρεσία προσπαθούμε να συνεργαστούμε με το Αφγανικό Κοινοβούλιο, να εκπαιδεύουμε κάποιους, κάποιο προσωπικό του Αφγανικού Κοινοβουλίου. Κροτές, εγώ πρόεδρε ζήτησα το λόγο για να σας τονίσω, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε διακοινοβουλευτική συνεργασία. Και θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία μας για την εισήγηση να μας στείλει περισσότερα στοιχεία, ούτως ώστε έτσι να έχουμε συνεχή ε, ενημέρωση. Να υπάρχει επομένως παρακολούθηση του τι γίνεται, τι, τι έργο επιτελείται, να γίνεται αξιολόγηση. Να μπορούμε να κάνουμε την αξιολόγηση όπως είπε ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε και ο κύριος Μίτσελ επίσης, παραταξιδεύουμε. Άρα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά τα ταξίδια, τις αποστολές που κάνουμε για να συναντήσουμε τους συναδέλφους από άλλα κοινοβούλια. Άλλωστε, αυτή η συνεργασία είναι στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της Επιτροπής μας. Και να έχει και μια συνέχεια. Άρα, να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και συνεργασία πάνω σε αυτό. Πρόεδρος. Και όσον αφορά την ε, κοινοβουλευτική συνέλευση της ΑΚΕ, έχω να σας πω ότι ε, με μέσω εκείνης μπορούμε να έχουμε συνεννόηση με τους ε, άλλους βουλευτές. Και συζητάμε τα κοινωνικά θέματα, θα πρέπει να έχουμε επίσης κάποιους εργαστήρια για να μπορούμε να συνεργαστούμε για κοινοβουλευτικά ζητήματα. Να οργανώνουμε ε, κάτι, κάτι σαν, σαν πρόβες εργασία. Ε, εργασίας. Ίσως πρέπει αυτό να τεθεί στο Προεδρείο της ΑΚΕ. Άλλες παρατηρήσεις. Κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική σας παρουσίαση. Θέλετε να δευτερολογήσετε συνοψίζοντας. Ναι, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια και την υποδοχή αυτή. Ναι, και, και από πλευράς IPU Πρέπει να σα πω ότι έχουμε εμεί περιορισμού στο έργο μα γιατί έχουμε προσωπικό μόλι 40 προσώπων. Ο κ. Κάσμαρ και μα είπε ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε περισσότερο τον κόσμο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Όσο γίνεται περισσότερο να ενημερώσουμε τα κοινοβουλία. Και όπως είπατε και εσείς, τα LDC θα πρέπει να είναι υψηλή προτεραιότητα και διαπιστώσαμε στο πρόγραμμα δράσης των Βρυξελών ότι πως θα δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν, να ακολουθήσουν οι ανεξόμενες χώρες. Ε, τους ενθαρρύνουμε τους, τους, τους, τους βουλευτές εκπροσώπους στο φορέα μας που είναι από τις τι ομένε χώρες να μας πούν τα, θέματα τους όσο γίνεται. Κύριε Γέλλερ, επίσης ε, συμφωνώ με αυτά που είπατε. Ναι, θα πρέπει το κοινοβούλιο να ασχοληθεί με αυτό το πρόγραμμα δράσης. Κατάλαβα τι είπατε όσον αφορά τις παρελήψεις που έχουν γίνει με την κυρία Άστον χθες τα είπατε. Για το ότι πολλές φορές αισθάνεστε ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις σας. Και αφού αυτό είναι διαπίστωση δική σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φανταστείτε πώς αισθάνονται οι βουλευτές των λιγότερων επιτυγμένων χωρών. Δηλαδή ο ρόλος είναι τελείως τυπικός, διακοσμητικός. ο κ. Μίτσελ μας είπε για τις ε, ε, ελλείψεις, ε, για το ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες υποστήριξη αποτελεσματική δουλειάς. Δεν έχουν, δεν έχουν τα μέσα στις χώρες εκείνες. Στη Σιέρα Λεόνα, ξέρετε, έχουν 124 βουλευτές και 10 υπαλλήλους για να εξυπηρετήσουν όλους για όλα. Φυσικά και δεν έχουν συνεργάτες, οι βουλευτές και, και με το ζόρι έχουν και, και συνδέσεις παροχή ίντερνετ για να δουλέψουν. με την Επιτροπή, με το Κοινοβούλιο, έχουμε διαρκή επαφή. συνεργαζόμαστε και σε επίπεδο ΠΟΕ. Είναι στενή η συνεργασία μας. Και συγκεκριμένα με τη δική σας ε, επιτροπή. Πάντως και πάλι να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε και μου δώσατε την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ. Επίσης ε, υποτίθεται ότι στην Τόχα θα συνεζητούνται και θέματα ανάπτυξης, τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, τόσο σημαντικό που ίσως δεν αρκούν μόνο μερικά λεπτά να το συζητήσουμε. Είναι το μέλλον της ε, πολιτικής της ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συζητούμε για πρώτη φορά, χωρίς έγγραφη επομένως με τον κύριο Γκέρνς μεγάλο γνώστη της υπόθεσης και άρα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής. Ο κύριος Μπέρναρτ, ο οποίο είναι διακεκριμένο μέλος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ασχολείται με τα θέματα αυτά, είναι παρόν και ως εκ τούτου Εάν θέλετε να ξεκινήσουμε, θα έλεγα εισαγωγικά ότι πρέπει να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής ώστε να επιφέρει ουσιαστικέ αλλαγές και να αξιοποιείται το πολιετές μέσων χρηματοδότησης 2011-2020 Χωρίς έγγραφο λοιπόν η πρώτη συζήτηση, ο κύριος Γκέρνης θα θυμάσει, αφού ακούσει τις απόψεις των συναδέλφων, ένα έγγραφο για την προσοχή μας συνεδρίαση. Σάρλ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητέ μου πρόεδρε. Όταν ε, μιλούμε για ατζέντα για την αλλαγή, τροποποίηση δηλαδή της, ε, του προγράμματος ε, για την ανάπτυξη, ε, πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα τι έχει αλλάξει. Έχουν, έχουν αλλάξει τα σύνορα. Είναι πιο ανοιχτά αλλά και πιο κλειστά. Είναι πιο ανοιχτά για τα προϊόντα, πιο κλειστά όμως γιατί δεν αφήνουν να περνάνε οι άνθρωποι. Το δεύτερο πράγμα που άλλαξε είναι το εύρος που έχει προσλάβει το διεθνές εμπόριο. Το διεθνές εμπόριο κινητήρας της παραγωγής πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο και χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία. Νομίζω ότι μιλάμε για 23 ε, εκατομμύρια δολάρια αύξηση του εσωτερικού του ακαθάριστου χώρου προϊόντος από το 2010, αλλά αυτό πάλι είναι ε, υποέλεγχο στοιχείο. Πλούτος λοιπόν που παράγεται τεράστιος, αλλά κακώ καταρρεπημένος. Ένα τρίτο πράγμα που αλλάζει είναι η σχέση μεταξύ των κρατών, συνέπεια της παγκοσμιοποίηση, όπως εξήγησαν νωρίτερα στην έκθεση για τη Λατινική Αμερική. Οι σχέσει λοιπόν μεταξύ κρατών αλλάζουν υπό την εξή έννοια ότι οι αποκλήσεις πλούτου μεταξύ κρατών μειώνονται, αλλά οι αποκλήσεις πλούτου στο εσωτερικό της κάθε χώρας ενισχύονται. Τέταρτο στοιχείο που τροποποιείται δεδομένα είναι η αδιάκοπη δυναμική στο παγκόσμιο, στην παγκόσμια κλίμακα δημογραφική δυναμική 6, έχουμε φτάσει πλέον στα 7 δισεκατομμύρια μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα και στα επόμενα έτη θα φτάσουμε πάρα πολύ γρήγορα στα 9 πράγμα το οποίο όμω δεν αναφέρουμε στα έγγραφά μα αρκετά συχνά. Κάτι άλλο που αλλάζει επίση είναι το κλίμα, οι κλιματικέ συνθήκε που οπωσδήποτε θα χαρακτηρίσουν τι συζητήσει μα για τι προσεχεί δεκαετίε. Έκτο σημαντικό σημείο αλλαγή, στοιχείο αλλαγή, είναι η φύση του ε, συστημικού κινδύνου που ενέχεται σε κάθε κρίση. Δηλαδή, μία πτώχευση τράπεζας ε, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου ή σε ελάχιστο χρόνο μπορεί να προξενήσει παγκόσμια οικονομική κρίση. Το 2008 είδαμε συνέπειες της πτώχευσης της Lehman Brothers που δεν περίμενε κανείς και τώρα μια τέτοια αντίστοιχη πτώχευση προξενεί κλειδονισμού σε κάθε τομέα, οικονομία, κοινωνικό, ακόμη και δημοκρατικά συστήματα μπορεί να αμφισβητήσει και να θέσει σε κίνδυνο μια τέτοια πτώχευση. Άλλο ζήτημα που αλλάζει είναι η ταχύτητα των τηλεπικοινωνιών. 8 στοιχείο αλλαγή. Όχι αρκετή και πάντω ε, όχι πάντα προ σωστή κατεύθυνση. Και η διαχείριση των παγκοσμίων, ε, της παγκόσμιας διακυβέρνησης με το G20, ένα νέο στοιχείο που είναι και ε, ευρύτερο αλλά και στενότερο. Ευρύτερο γιατί περιλαμβάνει ακόμη περισσότερα κράτη, αλλά παρόλα αυτά είναι στενότερο γιατί αποκλεί πάντα τα 80% του παγκόσμιου πληθυσμού, του πληθυσμού της γης, γιατί δεν, έχουν, δεν έχει αυτός ο πληθυσμός της γης επαρκές ΑΕΠ, ενώ έχει πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα που πρέπει να επιληθούν και τα οποία καλούνται κάποιοι άλλοι να επιλύσουν σε παγκόσμια κλίνικα, κλίμακα, πράγμα το οποίο βρίσκω παράδεκτο. Πάντως πρέπει να σημειώσουμε επίση τι σημαντικέ πρόοδους που υλοποιήθηκαν σε κάποιους τομείς, όπως πρόσβαση πρόσβαση σε φάρμακα. Πριν από 10 χρόνια, αν σας ε, έλεγε κανείς ότι το 2012 θα ήταν εκατομμύρια οι ασθενείς ανά τον κόσμο σε αναπτυσσόμενες χώρες που θα είχαν πρόσβαση σε αντιρετροϊκά φάρμακα, ε, θα σας παίρνανε για νερά ειδοπαρμένο. Όμως αυτή η ε, ιδέα που φαινόταν μάλλον ψευδέστηση στην εποχή εκείνη πριν από 10 χρόνια τώρα έχει καταστεί πραγματικότητα. Ένας άλλος παράγων αλλαγής είναι η εξωτερική δράση που βέβαια δεν είναι πάντα σαφής ε, ως προς ε, την δική μας τώρα των πραγματών. Δεν βλέπουμε ποιος έχει κάνει τι ακριβώς αλλά εν πάση περιπτώσει το έγγραφο που παρήχθη είναι καλό, αποτελεί μια καλή βάση συζήτησης και τα στοιχεία που έχουν αλλάξει νομίζω ότι βρίσκονται, ανέρχονται στο ύψο των προκλήσεων. Η βούληση, παραδείγματι, να επικεντρωθούμε περισσότερο σε κάποιου τομεί, συγκεκριμένου με σε μια ανεπτυσσόμενη χώρα, από πλευρά τη Ένωση τη Ευρωπαϊκής και συγκεκριμένα τρει τομεί, πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτοί οι τρει τομεί θα πρέπει όμω να ανταποκρίνονται στην πρωταρχική αυτή ε, κλίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιο χορηγού και δωρητή, ώστε να υποκαθιστά επιτυχώς αυτό που δεν μπορούν να πράξουν οι ε, μικρότερες κλίμακας εθνικοί παράγοντες και φορείς. Επίσης, σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε εδώ, να παραμείνουμε μέσα σε μια δυναμική προσέγγιση, σε μια προσέγγιση η οποία θα είναι σε θέση να επιφέρει αλλαγές, χωρίς όμως να αφισβητήσει το εξασφαλιστέν ήδη και εκτιμένο ε, λόγω υπερβαλλοντος ζήλου ενδεχομένω. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε σε επαγρύπνηση και υπογραμμίζω ότι στην Ευρώπη έχουμε δει αυτή την, ε, έχουμε αυτή την εμπειρία. Η πολιτική των μικρών βημάτων ήταν αυτή που έφερε τα αποτελέσματα. Γιατί αν στι αρχέ δεκαετία του 70 είχαμε προσπαθήσει να επιδιώξουμε το μέγιστο αποτέλεσμα, δεν είχαμε καταφέρει τίποτα. Και εδώ στα ανθρώπινα δικαιώματα, ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ενδογενέ και ε, αγκιστρωμένο στην εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το ξανασύσουμε μετά. Η κοινωνική ενσωμάτωση θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 20% τουλάχιστον της Ένωσης προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται και μια συζήτηση όπου η μάλλον προσεκτική διατύπωση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της Ένωσης με οδηγεί στο να διαπιστώνω ότι το τουλάχιστον 20% συνεπάγεται πόσο παραμένουμε σε ε, ποσά που μπορούν να ξεπεράσουν το 20% και ελπίζουμε ότι θα το ξεπεράσουν. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον το κεφάλαιο για την ε, ανάπτυξη, την ευρή ανάπτυξη που θα περιλαμβάνει στο των περισσότερου ε, στους κόλπους τους. Είναι πολύ καλή η διατύπωση, ανταποκρίνεται και στις δικές μου προσδοκίες, με προσεκτική η διατύπωση βέβαια. Και θεωρώ σημαντικό σε μία ε, συνεπή και συνεκτική προσέγγιση της πολιτικής ανάπτυξης να είμαστε προσεκτικοί και να συμπεριλάβουμε όλους τους παράγοντες της ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι με ιδιαίτερη ενάργεια το κεφάλαιο που αναφέρει την ανάπτυξη με μία συμπεριληπτική σφαιρική ε, προσέγγιση. Ε, στόχος δηλαδή είναι οι πόροι που διαθέτουμε να αποβαίνουν σε όφελος ολόκληρης της κοινωνίας και όχι ορισμένων. Αυτό πρέπει να προσδιοριστεί με πιο συγκεκριμένους όρους βέβαια στους, ε, στους κανόνες μας για την ανάπτυξη. Για τα δάνεια θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα αποτελέσουν μέσα και πρέπει να τα συζητήσουμε στο βαθμό που εξυπηρετούν τελολογικά τους σκοπούς που έχουμε προσδιορίσει. η υλοποίηση μέτρων που στόχο έχουν την άρση των ε, ε, δυσχεριών ή του ευάλωτου ορισμένων περιοχών ή χωρών της ανάπτυξης. Ναι, πρέπει βεβαίως να δούμε με βάση τις διαστάσεις της κάθε περίπτωσης ε, τι χρειάζεται, αλλά και με ιεράρχηση αυτών των διαστάσεων. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, από ό,τι διαπιστώνω, επιτακτική ανάγκη είναι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πιο αδύναμων. Αυτό θα πρέπει να έχει την προτεραιότητα εναντί του κάθε ζητήματο που θα κληθούμε να κρίνουμε. Έχει να κάνει και με τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί η καταπολέμηση της ε, φτώχειας είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Αν κάποιος δεν έχει να φάει μια μπουκιά ψωμί, δεν έχει καμία, κανένα δικαίωμα. Όποιο δεν έχει στέγη πάνω από το κεφάλι του, όποιο δεν έχει μια μπουκιά ψωμί, δεν έχει επιλογή παρά μόνο να πεθάνει ή να ψοφήσει, όπως έλεγε ένας ερευνητή της υπόθεσης αυτής, ε, μέσα σε μια γενικότερη αδιαφορία. Αυτό νομίζω ότι περιγράφει πολύ καλά ε, την ε, ιδιαίτερη προτεραιότητα και έμφαση που θα πρέπει να δοθεί στο δικαίωμα να απαλλαγεί κανείς από την φτώχεια και το οποίο πρέπει να υπερτερεί σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μέλημα η θέσπιση, το πλαίσιο ή η, ανα... κοινοποίηση αποτελεσμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ιδιαίτερα με εντυπωσίασε. Καθώς είναι ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα. Από η προσωπική μου πείρα γνωρίζω το γεγονό ότι δεν μιλάμε πολύ μεταξύ μα. Κάτι μέλη, Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση μπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήματα και χρόνια πριν είχα μιλήσει με τον Επιτροπούλτον για κάποια ζητήματα χρηματοδότησης ε, σε προγράμματα που είχε ο ίδιος καθοδηγήσει και είχαμε συζητήσει για το μέσον αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Εν προκειμένου η δημοσίευση αποτελεσμάτων έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση πιστεύω. Πρέπει νωρίτερα να ξεκινήσει ε, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου η προσέγγιση προς την, η δική μου η τοποθέτηση προς την προσέγγιση, η βελτιωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη που συζητούμε. Επίσης, διαβάστε τις προτάσεις της Επιτροπής, ε, επιτρέψτε μου να παρουσιάσω και εγώ τις δικές μου. Η έκθεση αυτή ε, τοποθετείται σε μια σειρά προτάσεων που έχουμε διατυπώσει και στο πλαίσιο της έκθεσης Κάτσμαρα και στο πλαίσιο μου εκθέσεως. Η έκθεση Κάτσμαρα περιγράφει κάθε στοιχείο τη ανάπτυξη. Εγώ νομίζω ότι εν προκειμένου θα πρέπει να περιοριστούμε σε κάποιε προτεραιότητε ή πάνω απ' όλα να προσδιορίσουμε ποιε είναι οι προτεραιότητες μα. Και θα σα καλέσω να ε, τοποθετηθείτε ω προς την εξή θέση. Εγώ λέω ότι πρέπει να είναι πολύ σύντομο το ψήφισμα, να υπογραμμίζει τις κύριες προτεραιότητες να προβάλλει τα κύρια σημεία, τα σημεία στα οποία χρειάζεται εμβάθυνση, τα στοιχεία εκείνα δηλαδή που θα είναι η δουλειά μας τα επόμενα χρόνια και θα κάνω συγκεκριμένα επτά προτάσεις ε, για τις οποίες θα ήθελα τις τοποθετήσεις σας. Για τις προτεραιότητες δηλαδή. Αυτά όλα που σας λέω δεν είναι ακόμη διαρθρωμένα και παγιωμένα, γιατί βεβαίω. Ε, θέλω να έχουν στον ευρύτερο πεδίο έκφρασης ε, οι συνάδελφοι. Πρώτη πρόταση λοιπόν. Με, την, ε, με αφετηρία την εξή διαπίστωση. Από όλου του παράγοντε ε, τη ανάπτυξη διαπιστώνουμε ότι ουδή είναι ε, τέλειο. Πλην όμω όλα αυτά που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω και διαπιστώνω ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από οτιδήποτε άλλο έχει τελεστεί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε την τεχνογνωσία, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να καταστήσουμε και γνωστό το τι έχουμε τεχνογνωσία αυτή. Πώ λοιπόν θα το καταφέρουμε αυτό. Ε, Χθε η συζήτηση με την ε, Λέβη Άστον μου επέτρεψε να εκφράσω τις θέσεις μου. Μου απάντησε η Λέβη Άστον ότι την απασχολούσαν ε, τα ίδια ερωτηματικά που είχα εκφράσει και εγώ, αλλά ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί το έργο. Πρέπει όμως το έργο αυτό να ολοκληρωθεί, να κλείσει το, έργο το εργοτάξιο και οι αρχιτέκτονες αυτού του εργοταξίου να μας πούνε εν τέλει ποια μορφή θα πάρει το σπίτι όταν θα έχει πλέον ολοκληρωθεί το έργο και παραδοθεί. Πρέπει πια να ξεκαθαρίσει η εικόνα. Μέχρι στιγμής είμαστε σε μια κατάσταση μάλλον ενηγματική και μόλις προσπαθούμε να εξίσουμε αυτή την λία, τόσο λία επιφάνεια, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν στοιχεία ερεθισμού, υπάρχουν προσδοκίες ε, αμφωτέρωθεν που δεν εκφράζονται, δεν είναι δυνατόν να εκφραστούν. Έρχονται άνθρωποι να μας μιλήσουν στην Επιτροπή μας οι οποίοι μερικέ φορέ, ε, βασιλικότερο του βασιλείου προσπαθούν να παραμείνουν και σιωπηλοί για να μην ενοχλήσουν σε ορισμένα θέματα και ω εκ τούτου εγώ θα πρότεινα να γίνονται συζητήσει τέτοιου τύπου και κλεισμένων των θυρών ώστε ο καθένα να μπορεί να μιλάει για τα προβλήματα πραγματικά τον απασχολούν ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση αυτού του ευρωπαϊκού αρχιτεκτονήματος της ανάπτυξης. Και νομίζω ότι και στα μέλη της επιτροπή μα, επιτροπή που είναι ανοιχτή, στην οποία ο καθένα μπορεί να εκφέρει τη γνώμη του, θα πρέπει να επισημάνουμε αυτή τη διάσταση. Ότι είναι ανοιχτή ακριβώ. Η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, η Κομισιόν, η Επιτροπή, πρέπει, ε, το Συμβούλιο πρέπει να είναι παρόντε. Για την απουσία δε του Συμβουλίου, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και άλλη φορά, είναι απαράδεκτο. Το Συμβούλιο καθεξάμεινο μόνο και για τρει μόνο ώρε συνεδριάζει με συμμετοχή δύο, τριών, τεσσάρων υπουργών και αν αυτό αποτελεί πολιτικό διάλογο μεταξύ κρατών μιλών, θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει στο έσχατο σημείο της πολιτικής ασυνέπειας και ε, απουσίας συνοχής. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξουμε μια πολιτική συνοχής που να εκφράζει τους 28 παράγοντες της ανάπτυξης ε, που εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της. Για το η φτώχεια, οι που έχουμε με μέρους θεσμικού εταίρους, πιστεύω ότι ή μη τι άλλο θα έπρεπε να μας επιτρέψει να φτάσουμε σε μια συνένεση ως προς μια ενιαία τοποθέτηση για την ανάπτυξη που έχει υπογράψει το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι όροι που χτίστηκαν μέσα σε συγκεκριμένε συνθήκες μπορούν ακόμη και να αποδομηθούν σε άλλες συγκεκριμένε συνθήκες. Εάν λοιπόν ε, οι τρεις εκείνοι οι οποίοι μπορούν, ε, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν αυτά που πρέπει να αλλάξουν, δεν είναι σε θέση να μαζευτούν σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν, τότε ίσως το Κοινοβούλιο πρέπει να μονομερώς να αλλάξει τα πράγματα, αφού αυτοί οι δύο-τρεις δεν μπορούν να βρεθούν στο Συμβούλιο. Έστω και αν τα λέμε χονδροειδώς, νομίζω ότι είναι εύστοχη περιγραφή. Η, ε, το έγγραφο επίσης υπογραμμίζει την ε, προσέγγιση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να εκδηλώνεται σε κάθε χώρο συζητήσεως, σε κάθε διάβημα που σχετίζεται με την ανάπτυξη ανά τον κόσμο. Και εγώ προσωπικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριο χορηγό, μεγαλύτερο χορηγό στον κόσμο, απαιτώ να συνενωθούν οι παράγοντες για να συζητήσουν το phasing out και τις νέες ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβει ο κάθε παράγον της ανάπτυξης. Όλοι αυτοί δηλαδή οι οποίοι πλέον δεν βρίσκονται σε συνθήκες ανάγκης αλλά έχουν τη δυνατότητα πλέον να δανείσουν χρήματα. 1,3 δις που δανείζει η Κίνα ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε για λόγους χρηματοδότησης ε, χρέους νομίζω ότι το ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ δεν νομίζω πρέπει να κάνουμε μια διεθνή οικονομική διάσκεψη για το θέμα αυτό. Όχι, πολύ συγκεκριμένου όρου με πολύ συγκεκριμένα κεφάλαια και θέματα για το ποιο θα πρέπει να συμμετάσχει σε θα πρέπει να χορηγήσει μάλλον, να δωρεί σε αυτό το νέο πλούτο που αναπτύσσεται. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ε, των αγράφων αυτών είναι οι προτάσεις Επιτροπής για καλή συνεργασία. Βεβαίως πρέπει να έχουμε πολύ προσεκτική προσέγγιση, παιδαγωγική προσέγγιση και εταιρική σχέση. Επομένως να δώσουμε χρόνο εφόσον χρειάζεται στις ε, σχέσεις αυτές για να προχωρήσουν. Ένα άλλο σημείο το οποίο δεν έχει καταγραφεί, δεν ξέρω γιατί, είναι το σχετικό με την ε, με, την, με το δημογραφικό, με τα ποσοστά των γεννήσεων. Νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρουμε όσο και αν δεν φαίνεται αρεστό και να καλέσουμε τον καθέναν να αναλάβει τις ευθύνες του. Πιστεύω ότι υπάρχουν στρατηγικοί εταίροι που μπορούν να πράξουν σημαντικό έργο ε, όπως η παραδείγματι το Ταμείο των Εθνών για το πληθυσμό, το οποίο το έχουν οικοτάρει οι για αρκετά χρόνια στην συγκεκριμένη περίοδο, όπου ε, Ε, προσχηματικά και λέγοντας ότι επειδή χρηματοδοτεί ε, δήθεν αμβλώσεις στην Κίνα ε, απέριπταν τη χρηματοδότηση αυτού του μέσου και ότι δεν ήταν αλήθεια ότι συμμετείχε σε αμβλώσεις, σε προγράμματα αμβλώσεων. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, έστω και αν έχει περιορισμένου πόρους και νομίζω εν προκειμένου ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί προς την επιλογή των στρατηγικών εταίρων τέταρτη σειρά προτάσεων. Θα πρέπει πιστεύω να είμαστε πολύ ψηφτικοί επίσης προς την απέτηση ειλικρίνειας κατά την διατύπωση και παρουσίαση των λογαριασμών. Αν δούμε λοιπόν τα ποσά τα οποία αφιερώνονται στην ανάπτυξη, είναι πολύ εντυπωσιακά τα στοιχεία. Δηλαδή κάθε, ε, κάθε ε, διαγραφή χρέους θα μπορούσε να ε, είναι δικαιούχο για χρηματοδότηση ε, με όρους ανάπτυξης. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε διακρίσεις, διότι χρέος το οποίο προξενείται επειδή γέμισαν οι τσέπε κάποιων δικτατόρων είναι άλλο από το χρέος το οποίο ε, δημιουργήθηκε επειδή βοήθησε στο να έχει καλύτερες συνθήκες και ευημερία ο λαό. Εάν λοιπόν ε, χρηματοδοτούμε σε όρους ανάπτυξης. Το χρέος το οποίο έχει πάει, ε, προέρχεται από ποσά τα οποία μπήκαν στις έπαιρες των δικτατόρων, τότε έχουμε κάνει μεγάλο λάθος. Και διαμαρτύρομαι διότι κάθε φορά που μιλάμε για διαγραφή χρέους βλέπουμε παράλληλα αύξηση της αναπτυξιακής βοήθειας που δεν είναι καμία ουσιαστική ε, βελτίωση της κατάστασης αλλά μόνο ε, προσχηματική. Επίσης, στου συναδέλφου, θέλω να αναφέρω ιδιαίτερα την υπαγωγή σε όρους, την ανέφερα νωρίτερα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, θα πρέπει να είναι ουσιαστική αυτή η υπαγωγή σε όρους μέσα σε μια δυναμική προσέγγιση, η οποία θα διαπιστώνει από πού ξεκινάμε και πού πρέπει να φτάσουμε και ε, Ποιου όρου ε, θα πρέπει να ορίσουμε μέσα σε μια εταιρική σχέση ειλικρινή, ανοιχτή, ώστε να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είναι απαραίτητο πιστεύω να συζητήσουμε το θέμα αυτό, να συνεννοηθούμε στο θέμα αυτό. Γιατί στα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσαμε να κάνουμε κακό με δύο τρόπους. Είτε μη διατυπώνοντας ερωτήσεις, είτε διατυπώνοντας όρους υπερβολικούς. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή στην υπόθεση αυτή, την ε, χρυσή ισορροπία και βεβαίως αυτό θα το εξασφαλίσουμε ακούγοντας τους ειδικού, εκείνους που έχουν την περισσότερη εμπειρία στην υπόθεση αυτή. Ένα έργο μάλλον ε, λεπτό και ευαίσθητο της διεθνούς διπλωματίας. Επίσης με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συμπληρωματικότητα όλων των ε, εταίρων, το είχα πει και νωρίτερα. για να πω ότι όταν μια χώρα αναπτύσσει εταιρικέ σχέσεις ε, με μια χώρα του Νότου Φερρυπίν, θα πρέπει, όπως λένε οι υπεύθυνοι της Επιτροπής, να προσκαλεί και τους λοιπού χορηγού Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λοιπά κράτη-μέλη Φερρυπίν. Θα πρέπει να λογοδοτεί Ως προς τα αποτελέσματα, μια και το ε, είπαμε νωρίτερα για την αρχική προσέγγιση αυτή η πληρωματικότητα μεταξύ παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπόν θεσμικών εταίρων και παραγόντων, πώς σκοπεύετε να την αναπτύξετε. Ιδέες δεν έχω. Συγκεκριμένω όμως εσείς ε, που καθημερινά στην εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών βλέπετε τις συνθήκες, ίσως έχετε τις σωστές, τις ουσιαστικές λύσεις. Ολοκληρώνω. Κάτι αναλύσει και τις προτάσεις μου, λέγοντας ότι είμαι θετικό απέναντι στο έγγραφο, στα έγγραφα που μας παρουσίασαν οι υπεύθυνοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα όμως διατυπώνοντας και την απέτηση να αλλάξουμε συμπεριφορές στο Ευρωπαϊκό Πούλ Ανάπτυξης το λέω αυτό έτσι διότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα όπως έχουν. Θέλουμε να αλλάξουμε την ανάπτυξη στον κόσμο. Πρέπει όμως η αλλαγή να ξεκινήσει από εμά πρώτα. Πρέπει να βελτιώσουμε τις αμοιβές σχέσεις σε σχέση με τα όσα αντιμετωπίζουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γκόρεντζ. είναι πάρα πολύ σημαντικό το, το, πόσο ωραία τα σκεφτήκατε όλα, πόσο πώς, πώς ενδιαφέροντα μας είπατε. Ε, φάνταστα, ε, όλα αυτά πρέπει να τα, προβλημα, να, τα, να τα συζητήσουμε. Ναι, θα πρέπει να συζητήσουμε, να, να απευθυνθούμε και προς Συμβουλίο και προς ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τα πάρουν όλοι ζεστά Επίση, συγκεκριμένα θέλουμε να γίνει μια κεκλεισμένων θυρών συνάντηση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί και μετά μια δημοσία συνεδρίαση να έχουμε και το Συμβούλιο και τριμερός να τα πούμε. Δεν θέλω κάποιος από τους να έχει την ε, και την εντύπωση ότι δεν τον αφήνουμε κάποιον ε, απ' έξω. Νομίζω ότι το, πιο σωστό είναι να τα συζητήσουμε όλοι μαζί. Chatham House rules, as um, which uh, enables us to talk very freely. Ε, ναι, θα πρέπει να γίνει σωστό υπό συνθήκε που να μπορεί ο καθένα να μιλά ελεύθερα. Έχουν τώρα την ε, εταιρική σχέση Κίνα-ΣΥΠΑ, 3,3 δίνουν οι, δίνουν οι Κινέζοι, δανείζουν στους Αμερικανούς, αλλά οι, Αμερικανοί με τις επενδύσεις τους δημιουργούν θέσεις εργασίας. Για φανταστείτε να δανείσουμε στην Ινδία ένα τρεις ε, υπό τον όρο ότι θα έχουν αλλακτικές μορφές ενέργειας και και θα μας δώσουν εμάς ε, την, την ευκαιρία για επενδύσεις. Φανταστείτε. Ηλεκτρισμό σε κάθε χωριό στην τέλος πάντων. Όλα αυτά είναι πολιτική ανάπτυξη. Ο κύριος Λάστρα. En primer lugar, quisiera agradecer al señor presentación. En esta ocasión eh, hablaré por... Ευχαριστώ τον κύριο Κέρενς για την εισήγησή του. Και επίση ο κύριο Κάσμαν μου είπε να τον αντικαταστήσω που είναι ο σχεδόν συγκεκριτής και να σα πω τη σκέψη του. Eh, πρώτα πρώτα. Να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον πίτροπο Πίμπαλτ για την για την διαβούλευση που ξεκίνησε το 2010 και έχουμε επίσης το πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε τη διαφορά. Το 2005 πρώτη φορά τα συμφωνήσαμε και είπαμε ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια να βασιστούμε στη συνθήκη της Λισαβόνας γι' αυτό και τέτοια πολιτική ανάπτυξη θεωρητική πολιτική μας ομάδα είναι πολύ ε, σημαντική. En este, en este primer lugar, ese perfil más alto, Αυτή η ανάδειξη που θα πρέπει να γίνει για, που, που έχουμε τις αμπροτεραιότητες ανθρωπινά δικαιώματα και την σωστή διακυβέρνηση πάντα με την αιρεσιμότητα. Ανάπτυξη. Η ανάπτυξη με εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, να δούμε τι γίνεται με, με την ε, διαφοροποιημένη αρρωγή, βοήθεια που θέλουμε να δώσουμε. Επίσης, να έχουμε περισσότερο συντονισμό και συνεργασία Ευρωπαϊκής και Κρατών Μελών και έτσι να πάμε σε μια πιο συνεκτική αναπτυξιακή πολιτική. Έτσι να πιάσει τόπο η πολιτική ε, συνεργασίας, αναπτυξιακή συνεργασίας που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ και δίνω το στην κυρία Κέλλερ. This um, thing about the in-camera meeting, maybe can because I mean usually if you exclude the public that sort of needs a justification. Σε σχέση με αυτή την συνεδρίαση και κλεισμένων, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα σε ανοιχτή συνεδρίαση να μιλώ ελεύθερα. Να σα πω κάτι άλλο από την προηγούμενη εμπειρία μου. Δεν θυμάμαι και συνεδριάσει και κλεισμένων στι οποίε η Κομισιόν να μίλαγε με περισσότερη ειλικρίνεια, πιο ελεύθερα τέλο Τώρα, όσον αφορά ε, αυτή την, την ατζέντα των αλλαγών, τη αλλαγή, ευχαριστούμε για τα καλά σα λόγια. Εμεί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστεί το, ο χαρακτήρα αυτού του εγγράφου. Γιατί χθε η Λέθη Άστον είπε ότι έχει χαρακτήρα συμπληρωματικό όσον αφορά την ε, συνένεση. Είπε όμως, τι είπε, τι για νόημα εδώ ακριβώς πώς το είπε, είπε ότι πρόκειται για το μέλλον της, ε, το μέλλον της ε, πολιτικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σχέση έχει επομένω ε, το, το έγγραφο αυτό, η ατζέντα τέλο πάντων, με την Ευρωπαϊκή Συνένεση. ανάπτυξη με εμπλοχή ιδιωτικού τομέα. Αυτό θέλουμε, ναι, αλλά για εμά, του πράσινου. η ανάπτυξη είναι μέσο επίτευξη. η οικονομική ανάπτυξη δηλαδή για να πετύχουμε την, την, ε, την, την, ανάπτυξη της, ε, μιας, ε, μιας χώρας. Η ανάπτυξη της οικονομίας είναι μέσο. Επομένως, πρέπει να θεωρήσουμε αυτές τις έννοιες εδώ, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε δει τι, θα πει αυτή η ευρεία η ανάπτυξη για όλους, πώς θα την πούμε, inclusive στα αγγλικά. Πρέπει να το, να το περιχαρακώσουμε αυτό. Ε, δηλαδή τι, να αγκαλιάσει όλα τα στόματα της κοινωνίας. Πολύ σημαντικό. Συζητήσαμε και με αφορμή τη Λατινική Αμερική. Είπαμε να μην γίνονται πλούσιοι πλουσιότεροι και φτωχοί φτωχότεροι. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε προς ε, έναν ορισμό, να βρούμε έναν ορισμό για το τι είναι αυτή η ανάπτυξη για όλους. Inclusive growth. Η χρηστή διακυβέρνηση, η ρησιμότητα. Για να δούμε. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Πώς συνδέονται όμως με τις παλαιότερες προτεραιότητες και την Ευρωπαϊκή Συνένεση, υγεία, περιβάλλον. Αυτά τώρα πώς θα, πώς, πώς θα ενταχθούν στην καινούργια πολιτική, θα τα αφήσουμε στην άκρη. Πώς θα άρουμε κάποιες αντιφάσεις που υπάρχουν, κάποιες συγκρούσεις. Πρέπει να έρθουν αυτές οι αντιφάσεις επομένω. Και ο κ. Πίμπαλτ επίση ε, μίλησε για την αιρεσιμότητα. Όχι, ποτέ δεν πρέπει να, να, να έχουν δασκαλίστικο ύφο. Έτσι θα το κάνει. Θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο προ τον συνομιλητή μα. Όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν σε αυτή την ε, ατζέντα για την αλλαγή. Επίση, εάν υπάρχει κάποιο γενικό κρατήρα έγγραφο θα πρέπει ίσως να δούμε τι είναι, ποια είναι η προσθεμένη αξία στα θέματα που μας απασχολούν. Η... Τίποτα δεν λέει πάνω σε αυτό η ατζέντα για την αλλαγή. Δεν φύγει τα αναψιακά θέματα που μας ενδιαφέρουν. Κρέμα. Θα πρέπει να το τονίζετε περισσότερο. Πώς εφαρμόζονται αυτές τις διακηρύξεις. Πώς θα έχουμε μεγαλύτερο συντονισμό, κοινό προγραμματισμό. Ε, να μπορούμε να πούμε έχουμε αυτό το στόχο. Εδώ έχουμε προσθέμενη αξία. Να, πώς διαρθρώνεται αυτή η ατζέντα για την αλλαγή. Άρα θα ξεκαθαρίσει όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω τίποτα από το ιδιωτικού τομέα και την εμπλοκή του. Αλλά όμως, Εντάξει, αυτό μπορούν να το κάνουν. Πάντα. Αλλά δεν θα μέσα χρηματοδοτήσουμε τον ιδιωτικό τομέα. Φυσικά και είναι σημαντική εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, αλλά δεν είναι το μόνο σημαντικό. Και ούτε ωφελούνται αναγκαστικά όλοι σε μια κοινωνία από την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα ρωτήσαμε κάποιο πράγματα τον Επίτροπο και δεν μας έδωσε απαντήσεις. Παρακαλούμε ομένω να μας ε, διαφωτίσει για όλα αυτά τα μυστήρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Κέλλερ. Κάποιους ορισμούς τους καθορίζει στον τομέα αυτό η Παγκόσμια Τράπεζα. Ο κύριος Κατσμάρεκ. Ε, E, Βασικά μπροστά μας θα έλεγα έχουμε μια εξαιρετική παρουσίαση του θέματος από τον κύριο, Γκέντς, ε, τον, Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί του σε κάτι. Δεν θα πρέπει να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε, θα ήθελα να πω ότι είμαι και εγώ υπέρ της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την Ανάπτυξη. Αυτό ήταν ένα επιτυχές βήμα στο οποίο είχε πάρει μέρος το Κοινοβούλιο. Και καταλαβαίνω και το δικαιολογημένο θα έλεγα του αιτήματο του κυρίου Γκέρενς για κεκλεισμένων των θερών συνάντηση. Πρέπει να συζητήσουμε με το Συμβούλιο και για να είμαστε έτοιμοι διαπραγματευτικά νομίζω ότι η κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση θα είναι χρήσιμη. Μπορούμε να εργαστούμε με τον ίδιο τρόπο λοιπόν όπως το είχαμε κάνει όταν προετοιμάζαμε την Ευρωπαϊκή Συνένεση. για την Κίνα τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει κανείς. Εγώ θα προτιμούσα ε, η Ρωσία φυσικά να μην βοηθάει την Συρία και η Ρωσία να μην διαφοροποιεί τις τιμές ε, φυσικού αερίου ε, ανάμεσα στην Ουκρανία από τη μία και τη Λευκορωσία από την άλλη. Αλλά η Ρωσία επηρεάζει με τον τρόπο αυτό αυτές τις χώρες οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από μας. Σχετικά τώρα με την αξιοπιστία των ε, στατιστικών στοιχείων και δεδομένων αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί τότε μόνο μπορούμε να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Δεν θα συμφωνήσω επίσης με μία παρατήρηση η οποία έγινε. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας πρώτα στη μείωση της φτώχειας και μετά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάποιες χώρες έφυγαν από την φτώχεια αλλά δεν έκαναν τίποτα ποτέ στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράδειγμα η Σαουδική Αραβία. Η εκρίζωση λοιπόν της φτώχειας δεν οδηγεί αυτόματα προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν αυτή την δράση να την προωθήσουμε παραλήλως. Ακόμα και σε περιοχές όπου η φτώχεια συνιστά ένα πολύ σημαντικό θέμα, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν το κάνουμε αυτό, τότε ίσως θα είναι πολύ αργά να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα αργότερα. Το θέματα λοιπόν που έχουμε μπροστά μας είναι δύσκολα, είναι θέματα τα οποία πολλές φορές προκαλούν διαφορετικού τύπου και αποκλίνουσες ερμηνείες και θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να προχωρήσει κανείς ε, για τα δημογραφικά στην Ευρώπη ε, που οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μια στάση απέναντι ε, στη δημογραφία και να μιλάμε με διαφορετικό τρόπο για το ίδιο θέμα για άλλες χώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα. Εμείς οι Ευρωπαίοι αυτό το οποίο θέλουμε είναι να ακολουθήσουμε κάποιες δημογραφικές εξελίξεις αλλά δεν θέλουμε τις ίδιες για άλλες χώρες. Περίεργο. Σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γκέρεν. Δυστυχώ με καθυστέρηση. Γιατί είχαμε ψηφοφορίε επί δύο ώρε στην Επιτροπή των Εξωτερικών. Έτσι συμβαίνει μια φορά. Κάποιε βασικέ ε, παρατηρήσει προ την ατζέντα για την αλλαγή. Νομίζω ότι έχουμε διαλέξει σωστό δρόμο. Κοιτάμε δηλαδή την βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων. Βεβαίω και χρειάζεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αναπτυξιακή πολιτική και μέσω την ατζέντα για τις, για τις για την αλλαγή μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Εδώ και καιρό ε, αγωνιζόμαστε για, μια, για ένα καλύτερο συντονισμό που δεν έχουμε επιτύχει απόλυτα γιατί δεν υπάρχει καλή ε, υλοποίηση των στόχων που ορίζουμε. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο και στα κράτη εκείνα τα οποία έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Χωρίς να λησμονήσουμε εκείνα που ανήκουν στο μέσο εισόδημα τα ε, little income countries. Με τα κράτη λοιπόν αυτά. Και αναφέρομαι, Φερρυπίν, στην Ινδία, η οποία έχει φιλόδοξο διαστημικό πρόγραμμα, αλλά ταυτόχρονα έχει και πρόβλημα πείνας αντίστοιχο με, τον, με τις χώρες. Πρέπει να αναπτύξουμε λοιπόν ένα λογικό διάλογο, ένα ουσιαστικό διάλογο και σε σχέση με τις χώρες ε, χαμηλού εισοδήματος να ε, αγωνιστούμε για την αποκατάσταση συστημάτων ε, κοινωνικών, υγειονομικής περίθαλψης που θα βελτιώνουν ουσιαστικά δηλαδή τις συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες. Έχουν δηλαδή ακόμη ε, πολλά να γίνουν και στα κράτη αυτά για την ανάπτυξη. Η χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία είναι αξίες που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερως. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκίξα στις προάλλες μας έλεγε ότι είναι παράδοξο να χρειάζεται κάποιος Αμερικανός να έρθει να μας, να μας αξιολογήσει την ε, αναπτυξιακή μας πολιτική. Αυτό νομίζω θα πρέπει να αποτελέσει ένα καλό μάθημα. Επίσης υπάρχει και η ε, κοινοποίηση μέσα από την ανακοίνωση του τι κάνουμε τελικά. Δηλαδή διαφάνεια, λογοδοσία, ορατότητα, όπως και συμμετοχή στις προσπάθειες. Παρακαλώ τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο για το θέμα αυτό. Θα ήθελα, δεν παρακολούθησα τον βιβλίο, σχετικά με τις κεκλεισμένο των θείων συνεδριάσεις. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι είμαστε, ε, θα έλεγα, ανώτερα όντα. Δεν είμαστε. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις συναντιόνται, ε, θα έλεγα, και κλεισμένα των θυρών, τα συνδικάτα επίσης, ε, η Επιτροπή. Αν θέλουμε το κάνουμε, αλλά το ότι όλοι θα πρέπει να είναι παρόντες στις συνεδριάσεις μας, όπου και αν είμαστε, δεν είναι αλήθεια εμείς κάνουμε εδώ τη δουλειά μας, αλλά για να προετοιμαστούμε χρειαζόμαστε ίσως να συναντηθούμε μόνοι μας. Ένα θέμα το οποίο έθεσε ο συνάδελφος και το οποίο δεν συζητάμε πολύ είναι το θέμα το δημογραφικό. Είχαμε κάποιους εδώ και λίγους μήνες δημοσιογράφους από την Ιρλανδία και είχαμε δει ότι η αύξηση του πληθυσμού το 50 θα είναι ε, πάνω από 2 δις. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να αγνοούμε. Από την άλλη δεν χρειάζεται να είναι κάτι το οποίο σχολιάζουμε και αναφέρουμε συνεχώς. Οι χώρες αυτές θα αποφασίσουν μόνες τους το τι θέλουν, τι είδους οικογένειες θέλουν, τι μεγέθη οικογενειακά επιθυμούν. Δεν θα τους πούμε εμείς. Δεν χρειάζεται λοιπόν εμείς να ασχοληθούμε με αυτό, πρέπει να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις. Σε αυτήν την Επιτροπή δυστυχώς και στο Κοινοβούλιο δυστυχώς καταψηφίσαμε μία τροπολογία να μην α, χρηματοδοτούμε κάποιες πολιτικές οι οποίες ε, οδηγούν στην δολοφονία because they are women, because they're female, gender side. So we do need a discussion on this. And even a liberal ε, πολιτικές οι οποίες επιτρέπουν τις αμβλώσεις. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε τις δολοφονίες αυτών των μικρών παιδιών. Λοιπόν, ε, τα θέματα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα, πρέπει να τα εξετάσουμε προσεκτικά. Πέρα από την πολιτική ορθότητα θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποιες, ε, κάποιο κοινό έδαφος, κάποιες κοινέ θέσεις και να βοηθήσουμε πραγματικά τον κόσμο να γνωρίζει ακριβώς ε, τι χρειάζεται να γίνει στον τομέα της αντισύλληψης κτλ. Δεν χρειάζεται καμία θεωρητική μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό. Πρέπει όμως ε, θα πρέπει να είμαστε κατά των αμβλώσεων, όλοι θα πρέπει να είμαστε κατά των φόνων των παιδιών, ανάλογα με το φύλλο κτλ. Ας, ε, αυτά είναι δεδομένα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μείνουμε σε αυτά στα οποία συμφωνούμε και ας δώσουμε την δυνατότητα σε όλες τις γυναίκες να μπορέσουν να προγραμματίσουν τις οικογένειές τους. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν και μέσω του Τσάρλς εδώ να έχουμε μια κοινή θέση. Μπορεί να έχουμε κάποιες διαφορετικές απόψεις, αλλά νομίζω ότι η βάση είναι κοινή για όλους και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε σε άλλους ιδέες που δεν είναι ξεκάθαρες και σε μας. Για πρώτη φορά στο DCI βάλαμε στόχους, είπαμε 30% στην βασική υγεία, 20% στην παιδεία, δεν ξέρουμε πώς θα το πετύχουμε αυτό. Και αν τυχόν υπάρξει μία αλλαγή το 10% σαν παράδειγμα στον τομέα της ε, εκπαίδευσης εννοούμε και τις υποδομές. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα πάνε τα πράγματα. Το θέμα είναι να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα. Η Κάφη Άστον μας είπε χθε ότι ο Πίμπαλξ εργάζεται σε αυτήν ακριβώς την ιδέα της, ε, της, της σχεδίασης, αν θέλετε, συγκεκριμένων μέτρων. Λοιπόν, το θέμα είναι σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είμαστε υπόλογοι για τις επιλογές μας. θα πρέπει μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξουμε σε μέτρα τα οποία να είναι απτά και κατανοητά και επιτεύξιμα. Ένα τρίτο θέμα. Αυτό που μίλαγα χτες η συνεκτικότητα. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα θέλετε ποτέ. Αν οι φορολογούμενοι ήξεραν ότι μετά από συνεργασία των εθνικών και των ευρωπαϊκών θεσμών θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα χρήματα που δαπανούμε στον αναπτυσσόμενο κόσμο όπου χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν καθημερινά ακόμα και σήμερα και θα μπορούσαμε τα χρήματα τα οποία να δώσουμε να αυξηθούν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής περίοδου και δεν το κάνουμε, αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο να ξεκινήσει μια κάποια πρωτοβουλία έτσι ώστε να συνεργαστούμε με τα κοινοβούλια των κρατών μελών για την μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στα κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούμε να φτάσουμε σε τεράστια ποσά. Να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο Bill Gates. Αν πετύχουμε το 0,30% τότε θα έχουμε πάρα πολλά χρήματα στη διάθεσή μας, θα φτάσουμε στα 30 δις για την καταπολέμηση της πείνας και αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις πολλές φορές και να συνεργαστούμε και να πάρουμε αποφάσεις και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Υπάρχουν πάρα πολλές προτεραιότητες στην επίσημη πολιτική μας και επειδή είναι πάρα πολλές οι προτεραιότητες δεν είναι πραγματικές προτεραιότητες. Θα πρέπει έστω να υπάρχουν κυλιόμενες προτεραιότητες. Επιτεύγματα σε κάποιους τομείς περνάμε σε κάποιους άλλους τομείς. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής αναδιοργάνωση ε, της σειράς και της ιεράρχησης των στόχων μας. Μόνο θα το πετύχουμε αυτό με έναν τρόπο αν ξέρουμε τους τρόπους με τους οποίους έχουμε πετύχει κάποιους στόχους ε, και αν ξέρουμε επίσης τους λόγους για τους οποίους κάποιους άλλους δεν τους έχουμε πετύχει. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στο μέλλον. Πρέπει να βελτιώσουμε και μπορούμε να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα και αυτά τα οποία είπε ο Τσάρλς σήμερα σίγουρα θα μας βοηθήσουν ιδιαίτερα. Ευχαριστώ κύριε Μίτσελ. Ξέρω ότι έχω εδώ δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να, τις ζητήσω, να τους ζητήσω να αποκριθούν στα σχόλια και τις ερωτήσεις που ε, έθεσαν τα μέλη της Επιτροπής μας. Μην αρχίσετε τώρα να διαβάσετε αυτά που ετοιμάσατε τις τελευταίες μέρες και μας κάνετε να βαρεθούμε. Αλλά προσπαθήστε να ανταποκριθείτε σε αυτά τα οποία ακούστηκαν σήμερα το πρωί έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και να είναι χρήσιμη η συνάντησή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Γκέρενς για μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για την ατζέντα για την αλλαγή. Πράγματι πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο προετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη στήριξη της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Δράσης. Για τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν λεπτομερώς θα σταθώ σε κάποια από αυτά. Καταρχάς η ατζέντα για την αλλαγή έχει σαν στόχο τον την προσαρμογή των προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής πολιτικής. Όπως είπε ο κ. Γκέρεντς, το παγκόσμιο πλαίσιο αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Συνένεση, απόψη μας είναι αυτή, παραμένει έγκυρη, παραμένει ενισχύ, ακόμα και αν υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να βελτιωθούν και να προσαρμοστούν αλλά επί της ουσίας οι στόχοι της, ε, και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Συνένεσης παραμένουν το έγγραφο πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμεθα να κινηθούμε. Δεύτερον, στα πλαίσια αυτής της αλλαγής πλαισίου θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Η οικονομική ανάπτυξη είναι αλήθεια ότι ε, τα τελευταία 9-10 χρόνια ήταν ιδιαίτερα υψηλή ακόμα και στις πολύ φτωχές χώρες. Αλλά η ανάπτυξη αυτή δεν μεταφράστηκε ουσιαστικά και αναλογικά με την βελτίωση των συνθήκων ζωής, με την μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη των δικτών που χαρακτηρίζουν το επίπεδο μιας κοινωνίας. Λοιπόν, η σημασία που πρέπει να, το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι η σημασία μιας ανάπτυξης η οποία να περιλαμβάνει τον άνθρωπο. Μιας ανάπτυξης στην οποία συμμετέχει η κοινωνία στο σύνολό της χωρίς αποκλεισμούς και αναφέρομαι εδώ και στους φτωχότερους της κάθε κοινωνίας στα σχέδια της παγκόσμιας, στους ορισμούς μάλλον της Παγκόσμιας Τράπεζας στις αναδιόμενες μεσαίες τάξεις όπως έτσι ε, σχεδιάζονται και προβλέπονται κάτι το οποίο θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς τους οποίους θα εξακολουθήσουμε βέβαια να είμαστε δραστήριοι γιατί η εκπαίδευση σαν παράδειγμα για θέματα υγείας και υγιεινής είναι προϋπόθεση mm για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ένα άλλο θέμα είναι η αύξηση των εταίρων που είναι παρόντες στα πλαίσια της βοήθειας για την ανάπτυξη. Ο κύριος Γκέρενς είπε ότι έχει μεγάλη σημασία να ξεκινήσει μια πιο διαρθρωμένη μορφή διαλόγου με αυτές που ονομάζουμε αναδυόμενες οικονομίες και που έχουν μια ευθύνη όλο και πιο μεγάλη σε σχέση με τη διεθνή ανάπτυξη και την κατανομή της ανάπτυξης αυτής. Αλλά θα έλεγα εδώ η ατζέντα για την αλλαγή δεν μας δίδει τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε, αλλάζει όμως κάποια πράγματα, ανοίγει κάποιους δρόμους σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα διαφοροποιηθούν οι εταιρικές μας σχέσεις με χώρες όπως τη Λατινική Αμερική Υπάρχουν πολλά τα οποία μένει να γίνουν ακόμα για να μπορέσουμε να ορίσουμε σωστά τις μεγάλες στρατηγικές μας προτεραιότητες στα πλαίσια των νέων μορφών συνεργασίας που θέλουμε να αναπτύξουμε με τις χώρες οι οποίες πιστεύουμε ότι έχουν περάσει σε ένα επίπεδο ανάπτυξης, δυναμικής ανάπτυξης που θα τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που έχουν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, προβλήματα φτώχειας, ανισότητας κτλ. Ένα άλλο σχόλιο για ένα από τα βασικά σημεία της ατζέντα για την αλλαγή, το θέμα της συγκέντρωσης των δυνάμεων. Φυσικά επί της αρχής συμφωνούμε. Πρακτικά όμως ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε αυτό. Εμείς σε αυτή τη φάση εργαζόμαστε για τις κατευθυντήριες γραμμές του προγραμματισμού των, και συνεργασίας των αντιπροσωπιών μας. Γνωρίζουμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνιμα καλείται να παρέμβει σε διάφορους τομείς και είναι πάρα πολύ δύσκολο να σεβαστούμε την αρχή της συγκέντρωσης των παρεμβάσεών μας. Είναι κάτι το οποίο θα αποτελεί μια πρόκληση. Να προσθέσω κάτι για το θέμα του συντονισμού. Η ατζέντα προτείνει ουσιαστικά δύο μέτρα Πρώτο μέτρο είναι η βελτίωση του διαλόγου και της κοινή αντιμετώπισης των, των αποτελεσμάτων στα πλαίσια της συνεργασίας κρατών μελών και επιτροπής. Και ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της, του κοινού προγραμματισμού δηλαδή κοινέ απαντήσεις κράτη-μέλη και Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη στρατηγική ανάπτυξη των διαφόρων χωρών. Και αν μου επιτρέπετε εδώ θα ήθελα Πρόεδρε να δώσω το λόγο στην συνάδελφο της, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ένα άλλο θέμα βέβαια στο οποίο θέλω να αναφερθώ και το οποίο θέσατε εσείς και το οποίο νομίζω ότι αξίζει να συζητηθεί είναι το θέμα της προτεραιότητας η οποία θα πρέπει να δοθεί στα θέματα της διακυβέρνησης. Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκδημοκρατισμός, δημόσια διοίκηση, δημοσια... Ε, ε, φορολογικές ρυθμίσεις. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά μια σωστής ατζέντα για την αλλαγή, η οποία δείχνει ότι θέλουμε να δημιουργούμε κίνητρα είναι στη φύση της αναπτυξιακής πολιτικής να δίνουμε κίνητρα για αλλαγές, κίνητρα για μεταρρυθμίσεις, να στηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές και όχι τόσο να στοχεύουμε από μόνοι μας να δημιουργούμε μια υπερβολική πολιτική αιρεσιμότητας μέσω προϋποθέσεων και γι' αυτό μας ενδιαφέρει πολύ και ε, η συζήτηση που γίνεται για τον τρόπο με τον οποίο ε, θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της δημοσιοποίησης των μέτρων που παίρνουμε στην ανάπτυξη διατηρώντας πάντα όλες τις δυνατότητες παρέμβασης τις οποίες έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Μωρό. Ο κύριος Χερνάντε Σόου έχει το λόγο από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην ε, Επιτροπή σας. Λέμε Φερνάντε Σόου και είμαι επικεφαλής της Υπηρεσίας για την ε, αντιξιακή συνεργασία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Είμαι διπλωμάτης, Ισπανός δούλευα στην ε, Ισπανική ε, μόνιμη αντιπροσωπεία πριν λάβω επομένω αυτήν την ε, θέση που σας προανέφερα. Είναι ένα παράδοξο μόρφωμα η υπηρεσία μας. Εκεί συνεργαζόμαστε διάφοροι από πολύ διαφορετικό background. Προσπαθούμε επομένως να συνεργαστούμε σε σχέση με αυτό το σε αυτό το σκοπό ε, ε, ουσιαστικά πρόκειται για κάποιο είδου διαδικασία διαβούλευση, ΔΕΦΚΟ και η ΕΕΣ. ΔΕΦΚΟ έχει την προτεραιότητα. Υπάρχουν, λοιπόν, ε, υπάρχουν αυτοί οι κοινοί σκοποί για του οποίου δουλεύουμε, γίνεται ο συντονισμό. Και υπάρχει τέλο πάντων συναρμοδιότητα, συνυπευθυνότητα για να πετύχουν του στόχου μα. Άκουσα τι παρατηρήσει του κ. Γκέρενς για το ποιος κάνει τι στην ατζέντα για την αλλαγή και εμεί προσπαθούμε επομένω να πάρουμε τα καλύτερα στοιχεία από τους μεν και από τους δε συναρμόδιους. Επίση, άκουσα διάφορες παρατηρήσεις σε σχέση με το αν ισχύει ή όχι η ενωσιακή συνένεση και εμείς ακριβώς <laughs> το ίδιο αναρωτιόμασταν όταν ε, φτιάξαμε αυτό το έγγραφο. Όχι, θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα και θεωρήσαμε ότι ισχύουν ακόμα τα περιεχόμενα της ε, συνένεσης. Ναι, ο κόσμος έχει αλλάξει. Ε, τώρα υπάρχουν καινούργιοι παίκτες στην ε, Κακέρα. Στο Μπουσάν αυτό πρόκυψε. Αναδύονται χώρες. Πολλές χώρες ξεφεύγουν από τη φτώχεια. Ακριβώ αυτό επομένω θα πρέπει να μας απασχολήσει. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτές τις αλλαγέ, να συντονιστούμε, να διαφοροποιήσουμε την στρατηγική μας. Να τι θα πει η ατζέντα για την ε, αλλαγή. Όπω όλοι, προσπαθεί να βρει την ισορροπία, όπως ε, σε όλους τους τομείς της ζωής, μεταξύ της ε, ανάπτυξης για όλους και της δημοκρατίας των δικαιωμάτων κλπ. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και παντού. Πρέπει να επικεντρώσουμε, να εστιάσουμε τι προσπάθειέ μα. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρετούμαστε από τα συμπεράσματα της ε, ενωσιακή συνένεση. Πρέπει να είμαστε όμω επιλεκτικοί για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα, να πιάσουν τώρα προσπάθειέ μα τέλο πάντων για την ανάπτυξη, για τη βοήθεια των πιο φτωχών, για τις σχέσεις με τους εταίρους μας, σε σχέση πάντα με το πώς εκείνοι διαχειρίζονται τα της ανάπτυξής τους. Πάρα πολύ ενδιαφέρον τους παρατηρήσεις που άκουσα. Θα πρέπει όντως να δούμε πώς στο μέλλον όλα αυτά τα διαχειριστούμε. Ε, πώς αυτή η διαδικασία αναθεώρησης θα επιτελεστεί. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν είναι αφετηρία για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για ε, να πετύχουμε το στόχο μας της ατζέντας αλλαγής τελικά. Οπότε προσπαθήσαμε και θα συνεχίσουμε προσπαθούμε να ασχοληθούμε με τους τρεις εκείνους τομείς Βέβαια το θέμα είναι τι πολιτική στάση θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει ομένω να κάνουμε κάποιε επιλογέ. Μέχρι σήμερα κάναμε επιλογέ, ε, αλλά όχι τόσο δεσμευτικά. Τώρα θα πρέπει να είμαστε πραγματικά επιλεκτικοί. Θα πρέπει να διαλέξουμε εκείνου του τομεί εκεί που ε, υπάρχουν οι προτεραιότητε για του εταίρου μα. Εκεί που έχουμε την προσταμένη αξία, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, με του άλλου δωρητέ. Άρα θα πρέπει να προβούμε σε πολιτικές επιλογές. συντονισμός και προγραμματισμός. Δεν ξέρω πώς τα, τα καταφέρουμε, αλλά εμείς προσπαθούμε, καθόλου όσο γίνεται περισσότερο και στην ΙΑΙΑΣ ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δούμε πώς θα υπάρχει ένας κοινό προγραμματισμός για το άμεσο μέλλον. Είναι προτεραιότητα αυτή. Να τα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη και να δούμε σε ποιου τομεί ποιο θα κάνει τι, να γίνεται τέτοια κατανομή εργασιών για να μπορέσουμε να, έχουμε απόδοση στις προσπάθειέ μας. Νομίζουμε ότι αν όλοι κάτσουμε γύρω το ίδιο τραπέζι και συντονιστούμε, θα πιάσουμε τις μα μας στην πολιτική ανάπτυξη, αλλά και γενικότερα έτσι θα περάσει προ τα έξω το μήνυμα της ανάπτυξης, γιατί αυτό ακούω να λέτε και εδώ, ότι είμαστε ένα παράγον που έχει μεγάλη περιοριστική σκηνή και θα πρέπει ομένω να συνεχίσουμε σε κάθε επίπεδο να, να, να προβάλλουμε το μήνυμα μα όπω και ο κ. Μίτσελ. Επίση θα πρέπει να μπλέξουμε τα Εθνικά Κοινοβούλια γιατί αυτό πρέπει να βοηθήσει τη συνεννόηση με τα κράτη-μέλη. Βεβαίω και θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τα Εθνικά Κοινοβούλια ούτως ώστε να περάσει αυτή η ιδέα του να ενεργούμε από κοινού. Επομένω, θα γίνει αυτό ο κοινό προγραμματισμό. Άκουσα επίση το πώς θα προσαρμόσουμε τις προτεραιότητες μας στις προτεραιότητες και στον προγραμματισμό των ε, αναπτυσσομένων χωρών. Γι' αυτό είπαμε να έχουμε πλέον προσαρμογή στον κύκλο λειτουργία των προγραμμάτων των χωρών εκείνων και μην έχουμε αυτό, αυτή την, την επταετία που είχε μέχρι τώρα. Επομένω, συνεργασία με τι χώρε αυτέ για τη λήψη υπόψη των προτεραιοτήτων του. Όσον αφορά τη διαφοροποίηση, φεύγω και θα γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε διαφορετημένες εταιρικές σχέσεις, διότι αυτές οι χώρες εμπισόμενες με μεγάλη τους χαρά ξεφεύγουν από τη φτώχεια. Άρα και εμείς θα πρέπει να προσαρμόσουμε την αναπτυξική μας πολιτική. Και, όπως είπε η Λεβιάστον για κάποιες χώρες θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσταθίες μας, για κάποιες άλλες θα πρέπει να κάτσουμε και να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται και με το πώς μπορούν εκείνες οι χώρες να βοηθήσουν άλλες. Άρα πρόκειται για μια εξεγόντως πολιτική σχέση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ μεστά τα όσα μας είπατε, λέει ο Πρόεδρος, και επομένω τώρα η Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει σε μια συνεννόηση. ακριβώς το που ζητήκε ο για συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επομένω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε. Ε, να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο και να τα συζητήσουμε σε περισσότερο βάθος. Κύριε Σό, πάρα πολύ καλά μα βλέπετε και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμω ο χρόνος ε, πιέζει. Κύριε Κέλλερ, μας αναφέρατε ε, πρόσωπα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζεται κάποιο είδου ε, επικαιροποίηση αυτής της ευρωπαϊκής συνένεσης, του Κονσένσους. Δηλαδή, τι θα κάνετε, θα προσαρμόσετε το Κονσένσους ή θα προσαρμόσετε την ατζέντα στο Κονσένσους, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, ίσως ε, δεν ήμουν αρκετά σαφής. Εσείς έλεγα ότι ότι το κονσένσους συνεχίζει να ισχύει 100% να ρίξετε μια ματιά. Αυτά όλα που εκεί αναφέρονται έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τους στόχους. Οι στόχοι δηλαδή του παρελθόντος ισχύων. Καλά, έχουμε κάποιες λεπτομέρειες εκεί, αλλά όχι. Δεν θεωρούμε ότι απαιτείται απεικαιροποίηση του κονσένσου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος ε, Γκιόνες τώρα καλύτερα να συνοψίσει. Παρακαλώ γρήγορα όμως. Πάντα, πάντα είμαι σύντομος Πρόεδρε. Κύριε Κορτές, συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Κύριε Κέλλερ, για τη συνεδρίαση και κλεισμένων. Κάνουμε ανοιχτέ συνεδριάσει. Κάνουμε συνεδριάσει ε, που δεν απέδωσαν τίποτα. Αλλάξαμε ε, απόψη με την κυρία Λεγιάστον που μας είπε ότι Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει μια διαδρομή, μια δουλειά που συνεχίζεται και μας ευχήθηκε καλή επιτυχία. Για μένα αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται ακριβώ. Υπάρχει κάποια δυσκολία. Ε, υπάρχουν, ε, υπάρχουν πραγματικά γεγονότα τα οποία δημιουργούν δυσκολίες ή όχι. Γιατί ε, αυτή η δυσφορία που υπάρχει προς Επιτροπής δεν, δεν, δεν την τιμά. Θα πρέπει όλοι να συντονίζονται για να πετύχει το σκοπό και είπα όμως ότι μια που δεν αποδίδουν εκείνη τη συνεδριάση, να βρούμε ενό άλλου είδου συνεδριάση. Δεν λέω ότι είναι σίγουρο, αλλά είναι μια, μια προσπάθεια τόσο ώστε να μπορέσουμε να αποσπάσουμε κάποια πράγματα από κάποιου που μπροστά στι κάμερε δεν θέλουν να τοποθετούνται, να εκφράζονται. Μέχρι σήμερα οι ανοιχτέ συνεδριάσει δεν απέδωσαν ε, τίποτα. Θυμάστε ότι το έλεγε, το είχε διαπιστώσει και ο παλιό συνάδελφο Μπουρλόν Προσπαθούμε. Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε τις απόψεις για να πετύχουμε αυτόν τον τόσο ευγενή, τόσο επενετό μας στόχο. Ανάλογα το τι πετύχαμε στο παρελθόν. Τριμερός προσπαθούμε να τα βρούμε. Τα τρία θεσμικά όργανα. Γι' αυτό το κονσένσου για την ανάπτυξη. Οι τρεις συμπλεκόμενοι πια έχουν σταματήσει να συνεννοούνται. Είναι απαράδεκτη η στάση του Συμβουλίου σήμερα. Στην Κινσάσα είδατε τι έγινε. Δεν πήγε καν το Συμβούλιο. Κι αλλού. Και όταν έστειλαν κάποιον, η στάση τους ήταν τέτοια που μας έκανε ρεζίλη, που ήταν ντροπή. Άρα θα πρέπει να αρθεί αυτή η δυσάρεστη κατάσταση που υπάρχει, Δεν είναι δυνατόν όλα να αναβάλλονται παρόριστον. Όλα να πηγαίνουν στις καλένδες. Θα πρέπει επομένω όντω η ανάπτυξη να καλύπτει όσο γίνεται περισσότερο. Θα πρέπει να βοηθά ε, αυτού που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, του πιο αδύναμους τη κοινωνία. Αλλιώ δεν έχει νόημα η ανάπτυξη. Αυτή είναι η ευθύνη αυτών που ασχολούνται με την ανάπτυξη. Ότι εκεί οι πλούσιοι έχουν και αυτοί κάποιες ευθύνες. Επίσης, δεν θα πρέπει όλα να τα φορτώνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη-μέλη, υπάρχουν και άλλοι. Και άλλοι που θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν για τον ιδιωτικό τομέα. Τα ίδια σχέδια και εκεί. Έχει ευθύνη ο ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι ακαδημαϊκό το θέμα. Δεν είναι φιλοσοφικό. Εταιρικέ σχέσεις. Αυτή η ιδιοποίηση. Θα πρέπει, επί τη βάση αυτής της αρχής ιδιοποίηση, να συνεχίζονται προσπάθειες. Και έτσι να θεωρούν δική τους την πολιτική μας και οι εταίροι μας. οι ίδιοι να την ασκούν μαζί μας. Επίσης, δεν έχω κάνει καμία προπαγάνδα όσον αφορά την υποχρεωτικότητα των αμβλώσεων. Είπατε η κυρία Ομπάκ, η οποία ήταν η υπεύθυνη για τα δημογραφικά στο ΝΟΙΕ, είναι ε, από τη Σαουδική Αραβία και η οποία και στο Αφγανιστάν και αλλού προσπάθησε ε, να περάσει το θετικό μήνυμα ε, όμως με παράδειγμα τρόπο μας επιτέθηκε γιατί υπάρχουν γυναίκες αναπτυσσόμενες χώρες που λένε ότι δεν θέλουμε πια να φέρουμε στον κόσμο παιδιά τα οποία δεν τα θέλουμε. Και αυτό γιατί οι άντρε δεν σέβονται την αξιοπρέπειά μα, άρα θα πρέπει να τι ακούσουμε. Θα πρέπει να του δώσουμε κάποιε απαντήσει. είναι θέμα σεβασμού της γενικής αξιοπρέπειας. Περί αυτού πρόκειται. Για τις γεννήσεις έχουμε 2-3% δημογραφικής αύξησης και αν έχουμε επίσης 3% ανάπτυξη οικονομική, τότε 3% και 3% 0. Άρα φρενάρεται η ανάπτυξη. Επομένως, οι χώρες που έχουν δημογραφική τέτοια μεγάλη ανάπτυξη θα πρέπει να έχουν ακόμα μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Αλλιώς έχουμε στασιμότητα της οικονομίας. Κύριε Κάτσμαρεκ, με όλο σεβασμό στο πρόσωπό σας και την ε, εκτίμησή μου στο κείμενό σας, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ λεπτό όσον αφορά τις ε, τις γεννήσεις το δημογραφικό. Όμως, ακόμα και ένα λεπτό θέμα, ακόμα και τα δύσκολα θα πρέπει να τα συζητούμε. Ας είμαστε επομένως ειλικρινείς και να ξεπερνάμε τα στερεότυπα τα οποία μας διχάζουν. Γιατί τα στερεότυπα αυτά δεν βοηθούν στη συζήτηση του προβληματισμού. Εντάξει, έχετε δικές προσέγγιση, αλλά θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Σύμφωνα με τον κύριο Μίτσολ και μετά άλλα που είπατε εσεί κύριε Κάσμαρικ, η Επιτροπή νομίζω ότι επιτέλεσε αξιόλογο έργο. Ακόμα πρέπει να κάποια πράγματα, τα οποία και θα λάβω υπόψη. Τώρα κάπως πιέζομαι από το χρονοδιάγραμμα. Ε, θα έχουμε το Μάιο το Συμβούλιο, ε, οπότε επομένω μια αντίστοφη μέτρηση πολύ πιεστική αυτή. Παρακαλώ και μην, μην, ε, μην, μην, μην με παρεξήσει κανένα. Αν κάποιο συνοχλήθηκε, ζητάω συγγνώμη. Ο μόνο θύματα φιλία τραφαγέλου. <laughs> Δικό σα πρόβλημα. Σα ευχαριστούμε. και για τα όσα είπατε και για τη διάθεση για συνεργασία. Τώρα νομίζω μπορούμε να καλωσορίσουμε τον πρεσβευτή της Κένιας, τον εξοχόδοτο Κίτο Πακ και τον νέο επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας στην Κένια. Με χαρά βλέπουμε εδώ και τον κύριο Τζον Κόρη, συμπρόεδρο στη μεικτή Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Ησυχία παρακαλώ. The next item, Το επόμενο θέμα και τελευταίο στην ημερήσια διάταξη είναι η παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεω για τι εργασίε τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή που επισκέφθηκε τον Δεκέμβριο την ε, Κένια τον Οκτώβριο-Νοέμβριο μάλλον. Η κυρία Στρίφλερ λοιπόν, επικέφαλη τη αντιπροσωπείας δεν μπόρεσε να έρθει, Όμω ο κύριο Κόρτε λόπε μα είπε ότι θα την αντικαταστήσει εκείνο. Και ε, Έχω συνεργαστεί με διάφορες οργανώσεις, παραγωγών, βοηθήσει στην προετοιμασία της εκθέσεως και τώρα θα μας ε, κάνετε την παρουσίαση για να ολοκληρωθούν τα στοιχεία της εκθέσεως. τις οποίες έχετε πρώτα διατυπώσει ένα, θα διατυπώσετε πρώτα ένα σχέδιο εκθέσεως και μετά θα ολοκληρωθεί αυτό και θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο κείμενο προτάσεων για την αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων στην Αφρική. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, με μεγάλη μου χαρά να σας παρουσιάσω το σχέδιο της έκθεσης όπως ε, φασίστηκε τον ε, Νοέμβριο. Η κυρία Στίφλερ δεν μπορεί να έρθει σήμερα, οπότε θα σας το παρουσιάσω εγώ. Καλώς όρισαν οι πρόσωποι της ΕΛΕΚ. Να τους ακούσουμε, τι έχουν να πούν και έτσι θα εμπλουτιστεί σίγουρα η σημερινή μας συζήτηση. Επίσης, χαιρετίζουμε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Και ο κύριος Λόντεβικ από την υπηρεσία εκπροσώπησης μας στην ε, Κένια. Βοήθησε πάρα πολύ. Και την ΕΚΟ Και ο πρέσβης της ε, χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλαμε με αυτή την αποστολή να αξιολογήσουμε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε τι γίνεται όσον αφορά αυτήν την και χρόνια ανάγκη όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια στο κέρας της Αφρικής. Πρόκειται για τη Βόρεια Κένια. Εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη ξηρασία. Ε, εκεί η κύρια δραστηριότητα είναι η εκτινοτροφία, τρόφιμα, ε, ορδευτικά έργα προσπαθήσαμε να οργανώσουμε να δούμε πώς θα προλάβουμε τις ε, φυσικές καταστροφές ε, που προέρχονται και από τις ε, ξηρασίες. Πήγαμε και σε κάποιο χωριό και ασχολούνται πάρα πολλές ε, ε, ε μη κυβερνικές οργανώσεις ούτως ώστε να, να αντιμετωπιστεί αυτή η ξηρασία και να δούμε πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση και επίσης πώς θα βοηθήσουμε στις προστριβές που δημιουργούνται λόγω της α, ξηρασίας. Ήρθαμε σε επαφή με τις αρχές, με τον ε, Πρωθυπουργό, ε, με εκπρόσωπους των ε, Βοσκών πήγαμε στο Κοινοβούλιο συναντήσαμε εκπρόσωπους διεθνών οργανώσεων μη κυβερνητών οργανώσεων ε, που συμμετέχουν στην, στην ανθρωπιστική βοήθεια όσον αφορά την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών Τρισήμιση εκατομμύρια κενιατών έχουν πληγεί από αυτήν την διατροφική κρίση και οι πιο ευάλωτοι βέβαια είναι η πιο φτωχοί, είναι η βοσκοί και η γεωργοί ε, σε αυτές τις ε, ξερές περιοχές, τις ημιέρημες ε, που έχασαν τα κοπάδια τους επομένως το θέμα ήταν το αν, πώς θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει αυτές τις συνέπειες αυτή την κρίση εάν είχαν ληφθεί προηγουμένως κάποια μέτρα. Θα πρέπει να έχουν γίνει κάποιες επενδύσεις εκεί. Τα δύο τρίτα εκεί ζουν κάτω το κατόφλι της φτώχειας. 5% ε, κατά μέσο όρο ε, για, όλο το, για όλη τη χώρα αναλφαβητισμός μεγάλος, 10,5% των ανδρών και 2,5% μόνο των γυναικών μπορούν γνωρίζουν ανάγνωση. Ε, πάρα πολύ λίγη άσφαλτος υπάρχει. Ε, οι δρόμοι, το, το δίκτυο είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και επομένω ε, είμαστε βέβαιοι ότι, η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει τι ευθύνε τη, κάτι να κάνει για ε, να μπορέσει να να κάνει κάτι για αποτελέσματα της κρίσης και να προλάβει για τις επόμενες. Έχουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ε, θα πρέπει να, ο ρόλος τους να αποκτήσει θεσμικό χαρακτήρα και να συμμετάσχουν και στις υπηρεσίες υγείας, δηλαδή θα πρέπει η κυβέρνηση να επενδύσει όσον αφορά την προστασία ε, αυτών που μένουν εκεί για το εισόδημα των κατοίκων αυτής της περιοχής, σε, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Θα πρέπει να γίνει περισσότερη διαφοροποίηση εκεί της οικονομίας. Αλλά αυτό δεν γίνεται αν δεν γίνουν κάποιες ε, επενδύσεις ε, για τις βασικές υπηρεσίες. Η κυβέρνηση θα πρέπει να βοηθήσει λοιπόν, τον πληθυσμό εκεί, όμως ε, οι εντατικές καλλιέργειες μόνο στο 1% αυτών των γεών να, αναεφαρμοστεί. εφαρμοστεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Η, πάντως έχει μέλλον η οικονομία ε, που βασίζεται στην βοσκή των ζώων. Θα πρέπει όμως να υπάρξει υποστήριξη με κάποιες πολιτικές και με κάποιες επενδύσεις. Έτσι θα βοηθούν οι κτηνοτρόφοι. Να σας πω τώρα τις βασικές συστάσεις της αντιπροσωπείας που εντάσσονται στο κείμενο. Πρώτα-πρώτα, το βασικό θέμα της αντιπροσωπείας είναι ότι δεν πρόκειται εδώ για ε, ακραία ανθρωπιστική καταστροφή. Όμως θα πρέπει με διαφορετικά έργα, διαφορετικές κινήσεις να βοηθήσουμε ούτω ώστε να καλυφθούν εκεί οι πιο ευάλωτοι. Συντονισμός, να βοηθήσουν οι αρχές και έτσι να έχουμε κάποιες στρατηγικές μακρόπνες για να υπάρξει διατροφική ασφάλεια και να προλαμβάνονται τα αποτελέσματα της ξηρασίας. Και έτσι τα χειρότερα θα τα αποφεύγουν. να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες πολιτικές, κατάλληλα μέσα, ούτως ώστε να υπάρξουν κάποιες βιώσιμες πολιτικές, οι διεθνείς δωρητές όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει και αυτοί να στηρίξουν την προστασία του πληθυσμού εκεί και για να αποφεύγουμε την διατροφική κρίση θα πρέπει να έχουμε πιο αποδοτικές παρεμβάσεις. Χρειάζεται κατάλληλη και έγκαιρη ανταπόκριση. Οπότε, οπότε χρειάζονται τέτοια βοήθεια γιατί τώρα αργήσαμε. Και έτσι θα σωθούν ζωές. Θα σωθούν και περιουσίες. Τρίτον, οι δωρητές θα πρέπει επίσης να εστιάσουν στους βαθιέ τους χωρίς, χωρίς να μην υπάρχει χωρίς να αποστερούμε από τον ντόπιο πληθυσμό τις δυνατότητες οι ίδιοι να αναπτύσσουν τις, δραστηριο... τις δυνατότητες τους. Παρά τις συνδίκες λοιπόν της ξηρασίας, δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη και θα πρέπει επομένω να κάνουμε περισσότερα και προστασία προληπτική. Έχουμε τώρα κάποιες ανισότητες και πάρα πολύ σκληρά έπληξαν αυτές οι ανισότητες τον πληθυσμό εκείνης της περιοχής της Βόρειας Σκηνής. Άρα πρέπει να λάβουμε ξεκάθαρες αποφάσεις και να βοηθήσουμε με την επαρκή προοικοδότηση. Γιατί αλλιώς η επόμενη ξερασία θα έχει ακόμα μεγαλύτερες δυσμενείς συνέπειες. Μπορούμε και πρέπει να λάβουμε αυτόν τον ρόλο να βοηθήσουμε την κυβέρνηση. Μέσα από την αιρεσιμότητα να έχουμε την οικονομική υποστήριξη και θα πρέπει να αποσπάσουμε εγγυήσεις από την κυβέρνηση της χώρας για το ότι η, χώρα, η κυβέρνηση δεσμεύεται να βοηθήσει αυτές τις προσπάθειες. Ευχαριστώ κύριε Λάστρα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε και πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση της αντιπροσωπείας. Ας ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο του Ινστιτούτου για 7 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και καταρχάς ευχαριστώ που μας προσφέρετε την ευκαιρία να σας κάνουμε αυτή την παρουσίαση η οποία δεν είναι ορατή για τους ερμηνείς. Πρόκειται για μια παρουσίαση που αφορά το μέλλον των βοσκοτοπίων στην Αφρική. Ορισμένοι έξιμων ίσως έχετε υπόψη την εικόνα ότι χάνονται τα βοσκοτόπια, ότι αυτή η νομαδική μορφή ζωής δεν έχει μέλλον στην Αφρική και ότι πρέπει οι νομάδες βοσκοί ε, να εγκατασταθούν μόνιμα σε κάποια περιοχή. Ίσως συμφωνείτε λοιπόν με αυτή τη ζωφερή προοπτική και πρόβλεψη. Ωστόσο υπάρχει και μια άλλη ε, έποψη, λιγότερο γνωστή, ότι δηλαδή είναι πολύ ε, δυναμική η οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές. Φερρυπίν, στο κέρας της Αφρικής, οι συναλλαγές σε ζώα, σε ζωικό κεφάλαιο, ξεπερνούν το ένα δις δολάρια. Συναλλαγές οι οποίες δεν καταγράφονται σε επίσημες στατιστικές, αλλά είναι υπαρκτές. Επομένως, ανθεί το εμπόριο στο ζωικό κεφάλαιο. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι το μέλλον αυτής της νομαδικής μορφής ε, ε, κτηνοτροφίας εξαρτάται από τη δυνατότητα πρόσβασης στις γέες. Στις εποχές ε, όπου χρειάζεται και στην αξία των γεών. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει επαρκής πρόσβασιμότητα και κινητικότητα στι γέε, αλλά χαμηλή προσβασιμότητα σε αγορέ. μπορεί κανείς να συνεχίσει να είναι ζωοτρόφο, ε, κτηνοτρόφος ε, νομάς όπως λέμε. Πλην όμως υπάρχουν και πολλές δυνατότητες ε, για δεκαετίες, εξού και οι δυναμικές εξαγωγές που διαπιστώνουμε. Άρα λοιπόν η εμπορευματοποίηση αποτελεί ήδη μια πραγματικότητα. Βλέπουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν ε, επιλογές διαφορετικές για τις οικογένειες αυτές. που στέλνουν τα παιδιά τους ε, αλλού για να ε, βρουν διαφορετικές συνθήκες ζωής. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με ζητήματα που αφορούν την ανθρωπιστική ανταπόκριση σε προβλήματα. Ε, θα σας δώσω λοιπόν σύντομα δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Η περιοχή Σομάλη της Αιθιοπίας, που είναι βέβαια όμορφη της Σομαλίας. Έχει αυτή την παραδοσιακή μορφή κτηνοτροφίας, η οποία όμως είναι το χρόνο έχει προχωρήσει σε σοφέστατη εμπορευματιοποίηση και τώρα έχει δημιουργηθεί μια νέα τάξη κτηνοτρόφων ομάδων ευπορών που χρησιμοποιούν ε, και την κινητικότητα αυτή και τις γέρες τους για να εξάγουν τα προϊόντα τους, τα ζώα τους. Άρα ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια του συστήματος και τα καταφέρουν και τα καλά. Μετά έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που έγκαθαν τα σαστικά κέντρα, διαφοροποιούνται ως προς δραστηριότητε τους με επιχειρηματικότητα, με νέες επαγγελματικές δυνατότητες που μπορούν να συμπληρώσουν την παραδοσιακή μορφή της ε, νομαδικής κτηνοτροφίας και έχουμε και αυτούς που εγκαταλείπουν το σύστημα και οι οποίοι χάνουν την πηγή εισοδήματό τους και ε, αγωνίζονται για να βρουν εναλλακτικές πηγές ε, εσόδων. Αυτή είναι που χρειάζεται περισσότερο την ανθρωπιστική βοήθεια. Το καθοριστικό λοιπόν στοιχείο εδώ είναι η εμπορευματοποίηση που αποτελεί σημαντικό παράγοντα και κινητήριο μοχλό. Και σχετίζεται βέβαια με την ευρύτερη συζήτηση που είχατε και όταν ε, ήρθα εγώ στην αίθουσά σας, δηλαδή την ε, ε, ισότιμη ανάπτυξη. Ανάπτυξη υπάρχει στις χώρες αυτές που όμως δεν είναι ισότιμη και ισοδίκαια μοιρασμένη. Κάποιοι γίνονται πιο πλούσιοι ενώ κάποιοι άλλοι χάνουν το παιχνίδι και τον αγώνα δρόμου. Στο καρονόζι της Ουγκάντα τώρα, ένα άλλο παράδειγμα. Καθώς έχει περιοριστεί σημαντικά η πρόσβαση στη, στα βοσκοτόπια, στις γέες και παραμένουν ε, περιορίζεται η κοινομαδικότητα, η κινητικότητά τους δηλαδή, βλέπουμε ότι βρίσκουν διαφορετικές λύσεις προσπαθώντα να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει. Επομένω, το μέλλον αυτό, αυτή τη μοναδική μορφή κτηνοτροφία εξαρτάται από το ε, που βρίσκεται κανεί. Ε, πολλά διαφορετικά στοιχεία διαπιστώνονται σε διαφορετικέ ή χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι κάθε περιοχέ. Δεν υπάρχει ομοιογένεια δηλαδή μεταξύ των περιοχών των βοσκοτόπων. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε πολιτική και ανταπόκριση που θα δοθεί σε, στις συνθήκες αυτές πρέπει να είναι πολύ περίπλοκη. Πολλά πράγματα συμβαίνουν, νέα πράγματα συμβαίνουν σε διαφορετικές περιοχές. Επιπλέον αυτού, και χωρίς εκπλήξεις, εάν κοιτάξουμε τις εξελίξεις στη νομαδική κτηνοτροφία σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως Φερρυπίν, Βόρεια Αφρική ή Μέση Ανατολή, έχουν περάσει μέσα από τις ίδιες αυτές τις μεταλλαγές. Είτε προχώρησαν, επεκτάθηκαν, εμπορευματοποιήθηκαν, είτε εξαφανίστηκαν. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Αυτό που θέλετε να σας πω ασφαλώς είναι το ότι πρέπει να γίνει. Η Κρίσιμη, πιστεύω, του τελευταίου έτους εξέλιξη είναι η αναδυσή του πλαισίου χάραξη πολιτικής των κρατών της Αφρικής για τα βοσκοτόπια και την ε, νομαδική κτηνοτροφία στην Αφρική. Πρόκειται για μια πολιτική, ε, ένα πολιτικό πλαίσιο αφρικανικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς πρέπει να υποστηρίξει την ανάπτυξη και τη λειτουργία αυτού του πλαισίου με αρρωγή προσφορά δηλαδή των πόρων που χρειάζονται και ευαισθητοποίηση ως προς, το ως προς το περιεχόμενο αυτού του πλαισίου που θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην, Ευρωπαϊκή... στην Αφρικανική Ένωση και επίσης ε, πιο συγκεκριμένα ε, χώρες, ομάδες που ενσωματώνονται σε αυτό το πλαίσιο με τις σχετικές ε, προσαρμογές από πλευράς ευρωπαϊκής μπορούν να ε, δουν και την συγκεκριμένη ανταπόδοση. Το πλαίσιο λέει δύο πράγματα βασικά ως προς την ανταπόκριση του πρόγραμμα. Λέει υποστηρίζουμε τα, την ομαδική κτηνοτροφία ως ένα βιώσιμο μέσο εξοικονόμησης του των προστοζήν. Έχει δώσει, όπως είπα, πολύ καλά αποτελεσματαμένα δις συναλλαγές ε, σε ζωικό κεφάλαιο ε, μόνο στο κέρας της Αφρικής. Δεν υπάρχει κρίση εκεί. Αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να υποστηρίξουμε εναλλακτικέ ιδέες και μπορεί να έχει την επιλογή ε, ο ενδιαφερόμενος να μείνει μέσα στο σύστημα ή να βγει εκτός συστήματος. Τρίτη παρατήρηση. Υπάρχει το θέμα της εναρμόνισης των προγραμμάτων και των στρατηγικών ε, των ανθρωπιστικών και αυτών με τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν σαν στόχο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα εδώ και δεκαετίες. Ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, δεν εκπλήσεται κανείς, ξέρουμε τι περίπου θα συμβεί και πού θα συμβεί. Αλλά παρόλα αυτά η θεσμική θα έλεγα συνήθως απόκριση είναι μια απόκριση ε, έκπληξης και τέλος, το μέλλον είναι διαφορετικό ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξουν αναλύσεις ειδικέ για κάθε χώρα, οι οποίες να προσαρμόζουν τα θέματα τα τοπικά στο ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό σημαίνει συστηματική επανεξέταση των δεδομένων και όπου είναι δυνατόν την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Κάτι. Πριν δώσω τη δυνατότητα στον Φίλιπ να σχολιάσει, να επανέλθω σε αυτά που έλεγε ο Ρικάρντο. Αυτά τα οποία μόλις ακούσαμε, νομίζω ότι ταιριάζουν με τις παρατηρήσεις που κάνατε επί τόπου, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, σίγουρα. Κύριε Πρόεδρε, στην έκθεση ρητός αναφερόμαστε στην ομαδική κτηνοτροφία. Και επίσης έτσι είναι δυνατόν να διαπιστωθεί και στην αποστολή που κάναμε ε, το ότι μιλήσαμε με πολλούς από αυτούς τους κτηνοτρόφους και θεωρούμε ότι κατά κάποιο ότι πρόκειται τέλος πάντων για, για μια μεγάλη μακραίωνη εκεί παράδοση. τα είδαμε, τους, ξανα, τους ξαναείδαμε, τους ξαναείδαμε και μπορέσαμε τέλο πάντων έτσι να συλλέξουμε πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ό,τι έγινε. Κάναμε δουλειά. Και πιστεύω θα επηρεάσουμε σε εξελίξεις στην περιοχή. Επρόκειτο για την παραμεθόρια περιοχή, προς την Αιθιοπία, το Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις ε, δύο ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Διάβασα και τη γραπτή έκθεση. Είναι μια εξαιρετική έκθεση. Έκθεση η οποία περιλαμβάνει ένα περιγραφικό κομμάτι λεπτομερέστατο, περιλαμβάνει όμως ταυτόχρονα και σημαντικά συμπεράσματα και τα συμπεράσματα αυτά θα έλεγα θα μας είναι πολύ χρήσιμα όταν εργαστούμε ε, για το ψήφισμά μας, για την έκθεσή μας. Χαίρομαι επίσης και για το ότι η έκθεση αυτή συγκεντρώνεται στο θέμα ακριβώς της ελεύθερης βοσκής. Δύο είναι ε, τα στοιχεία τα οποία πρέπει να μην αγνοήσουμε εδώ. Ε, πρώτον, μία, ένα από τα βασικά στοιχεία της κρίσης είναι η περιθεριοποίηση και το μόνιμο έλλειμμα επενδύσεων στις α, ε, μη γόνιμες ε, περιοχές. Ε, παστερσκих 350 Στις ζώνες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ξηρασίας επίσης czy było w 2011 e, Μέχρι τώρα είχαμε τόσα θύματα όσα είχαμε και το 2011 λόγω των εθνοτικών συγκρούσεων. Και αυτό θα έλεγα εξηγεί το ενδιαφέρον που έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Τα δύο θέματα αυτά λοιπόν έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα. Η έκθεσή μας αναφέρεται σε μια γενική στήριξη της ελευθέρας βοσκής, της δραστηριότητας αυτής της οικονομικής, και αυτό το οποίο υπογραμμίζεται από τον δεύτερο εισηγητή είναι μια κατάσταση πιο αναλυτική που αναφέρεται σε πιθανά σενάρια γενικά ανάπτυξης ε, κάτι το οποίο δεν είναι αρνητικό, είναι συμπληρωματικά τα έγγραφα όπως είπα μεταξύ τους. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε τα δύο αυτά έγγραφα παράλληλα. Είναι δύο έγγραφα πολύ συγκεκριμένα και θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούν οι συνάδελφοι με τον σωστό τρόπο και να το θυμίσουμε αυτό και στους συναδέλφους που είναι απόντες σήμερα. Ευχαριστώ. Φίλιπ. Υπάρχουν και άλλα θέματα όπως η ειρηνευτική διαδικασία, οι πρωτοβουλίες του Κόφη Ανάνα, η φροντίδα φυσικά για την Ελευθέρα Βοσκή. Ο εκπρόσωπος σε πάση περιπτώσει αντιπροσωπείας μας στην Κένια έχει το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Τόρες Λάστρα για την έκθεση την οποία προετοίμασε δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να φανώ εδώ υπερβολικός, αλλά θα ήθελα να πω ότι πράγματι είναι κάτι το συμβατό σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε πει στο παρελθόν. Σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούμε να ελέγξουμε την κατάσταση, να την αξιολογήσουμε μετά από την πρόκληση των ζημιών από τις διάφορες καταστροφές. Και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κατσμάρεκ έχουν πολύ σημασία θα έλεγα και είναι συμβατά με το PDNA και τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Επιτροπή σας που για ιατρικούς λόγους δεν ήμουν παρόν όταν επισκέφθηκε το Ναϊρόμπι. Και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και τους κενιάτες ομολόγους μου. Ε, έχει σημασία και συνεχίζει να έχει σημασία να ανοιχνεύσει κανείς σε διαρθρωτικούς θα έλεγα τρόπους ε, ε, αντιμετώπισης της έλλειψης τροφίμων σε αυτό το κομμάτι της Αφρικής. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Υπάρχουν πολιτικοί λόγοι, υπάρχει το θέμα της περιθεριοποίησης των άγωνων γενικότερα εδαφών, Υπάρχει το θέμα της ανασφάλειας, ιδιαίτερα στο βόρειο-βορειοανατολικό κομμάτι της Κένιας, επηρεαζόμενη από την Σομαλία, μείωση των βροχοπτώσεων και πτώχευση ενός μεγάλου κομματιού του πληθυσμού. Για να προλάβει κανείς τέτοιου είδους καταστροφές Φυσικά δεν μπορεί κανείς ε, να αποφύγει την ξηρασία, αλλά μπορεί κατά κάποιο τρόπο να προγραμματίσει έτσι ώστε να αντιμετωπίσει καλύτερα τις συνέπειές της. Είναι λοιπόν ένα νέο θέμα εδώ μπροστά μας, το θέμα της στρατηγικής στο κέρας της Αφρικής. Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση στη Σομαλία, δεν θα παραπέμψω εδώ στο τι συνέβη στην διάσκεψη στην, στο Λονδίνο για τη Σομαλία. Ακούσαμε επίσης και τον Αλεξάνδερ Όντος, τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, πήγε για πρώτη φορά στην περιοχή ε, πριν από λίγες εβδομάδες. Important what Mr. Catley said, the future of pastoralism, commercialization. This is not a mean affair. Obviously it's up to the societies. Οι κοινωνίες λοιπόν και οι τοπικοί πληθυσμοί θα αποφασίσουν το τι επιθυμούν και εμείς θα προσπαθήσουμε να τους στηρίξουμε στις αποφάσεις τους αυτές. Δεν θα πούμε εμείς από εδώ το πώς θα πάνε τα πράγματα. Έχει μεγάλη σημασία να μην αγνοεί κανείς το πόσο γρήγορα αυξάνονται και οι πληθυσμοί στην περιοχή αυτή της Αφρικής. Την εποχή της ανεξαρτησίας το 1963 υπήρχαν 7 ε, εκατομμύρια κενιάτες. Σήμερα είναι 40 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο το χρόνο αυξάνονται και το 50 θα είναι 83 εκατομμύρια αν πάει έτσι η κατάσταση, κάτι το οποίο δεν μπορούμε φυσικά να πούμε ότι μπορεί να είναι εφικτό σε επίπεδο στήριξης του πληθυσμού αυτού και κάλυψης των αναγκών του. Παλεύουμε παρόλα αυτά να αντιμετωπίσουμε το θέμα μεσοπρόθεσμα με σωστό τρόπο. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε α, τις ανθρωπιστικές παρεμβάσεις ευαισθητοποιώντας και της εθνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης της Κένια έχει μεγάλη σημασία. Εμείς θα είμαστε εκεί για να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση αυτή είτε εμείς, είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε η ΕΚΟ συνεργαζόμαστε για να βοηθήσουμε. Είναι θετικό το ότι το Σύνταγμα του Κενιατικό και οι πολιτικές που ακολουθεί η Κένια αναγνωρίζουν τον ξεχωριστό ρόλο που έχει η δραστηριότητα της ελευθέρας βοσκής, ιδιαίτερα στις περιοχές που εν μέρει υποφέρουν από, από ξηρασία. Οι εξελίξεις, οι θεσμικές, οι οποίες μένει ακόμα να προχωρήσουν, βρίσκεται υποσυζήτηση η αποκέντρωση και η οικονομική διαχείριση από πλευρά των τοπικών αρχών των περιφερειών αυτών είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση και η εφαρμογή τους. Η κυβέρνηση της Κένια έχει δώσει 70 εκατομμύρια ευρώ το 2011-2012 για την ανάκαμψη από την ξηρασία, την εισαγωγή χωρίς φόρο αραβοσίτου,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 compliment the colleagues from ECHO for their efforts, because they've been quite considerable. Thank you very much, Chairman. Thank you, Your Excellency. It's good to hear that ECHO is anticipating disasters. Ότι το ΕΚΟ μπορεί να προλάβει ή τουλάχιστον να προβλέψει κάποιες από τις φυσικές καταστροφές. Η Επιτροπή παρακαλώ. Δύο λεπτά μόνο. Πρόεδρε, κανένα πρόβλημα. Και δύο και τρία. Πολλά. Καλά ακούσαμε και από την έκθεση του Κοινοβουλίου. Και θα ήθελα να συμφωνήσω με όλα τα θετικά σχόλια που ακούστηκαν για την αντιπροσωπεία στην Κένια. Όσον αφορά την ανάλυση των όσων συνέβησαν ε, στο κέρας Αφρικής πέρυσι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανάλυση ε, προσπαθούμε να επανενταχθούμε, να επαναδεσμευθούμε καλύτερα στη, και να γίνει πιο ορατή η παρουσία μας ε, στο κέρας Αφρικής και ως εκ τούτου υπ' αυτή την έννοια οι προτάσεις που ακούστηκαν σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πολλά από αυτά που ακούστηκαν συμφωνούν με τις αναλύσεις της Επιτροπής στο στάδιο αυτό. Τα ενδιαφέροντα ζητήματα που προτείνει ο εισηγητής μας αναγκάζουν να αναλογιστούμε σε ποια πρέπει να επικεντρωθούμε. Υπάρχει το ζήτημα της ε, εκλογή αλλά βέβαια αυτό περιορίζεται και από τους φυσικούς πόρους και από τις πιθανές ή μη εναλλακτικέ κτλ. Υπάρχουν ε, προϋποθέσεις που μπορούμε να ακολουθήσουμε και μία εναλλακτική είναι η ανάγκη για δίκτυα ασφαλεία και για μέτρα τα οποία πάνω απ' όλα θα λαμβάνουν υπόψη τι ανάγκε του πληθυσμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλετε να επανέλθετε παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλες σας τις παρατηρήσεις. Για τη βοήθεια τη γραμματείας που ήταν όπως πάντα πάρα πολύ πολύτιμη κατά την αποστολή. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι είχαμε μία συνάντηση εργασίας με την αντιπροσωπεία της Ένωσης στην Σομαλία. Τα είπαμε το χρόνο. Ε, μίλησαμε για τα προβλήματα της χώρας για τον Ναϊρόμπι και συζητήσαμε για το τι μπορεί να κάνει η ΑΚΟ για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή. Πάρα πολύ περίπου τα πράγματα. στη βοήθεια του στρατού, πώ είναι μέσα από τα λιμάνια της χώρας να, φτάσουν, φτάσει παντού η βοήθεια. Ε, Κένια, Σομαλία. Για μια τόσο περίπλοκη κατάσταση, μια τόσο περίπλοκη περιοχή. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το feedback που πήραμε. Και ήδη διαπιστώσουμε επίση ότι η αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί επιτελεί και σχετικό έργο. Ρικάρντο, ευχαριστώ. Είναι την προσωπία της χώρας. Ε, κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας ευχαριστήσω. Also want to Ευχαριστούμε και για την, την σας στον Αεροβία πάρα πολύ σημαντικά. Αυτά τα οποία έγιναν όσα και όσα επέδωσαν σήμερα εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικά. Διάβασα την έκθεση της Διακοινωτική Επιτροπής και φυσικά δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με όλα όσα ανεφέρθησαν. Κάτι γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και θίγει πάρα πολύ σημαντικά ουσιαστικά προβλήματα. Νομίζω ότι τα συμπεράσματά σας θα πρέπει να αποτελέσουν μια βάση ε, και έτσι να συνεχιστεί ε, η δουλειά που κάνουμε αντιμετωπιστεί ε, ο λοιμός στην χώρα. Βεβαίως ξέρουμε ότι άλλο ξηρασία και άλλο λοιμός θα πρέπει επομένω να αναζητηθούν λύσεις. Πάντως, όσον αφορά την έκθεση, θα πρέπει να σας πω είτε περάσει όλοι είτε όχι δεν συμφωνώ με το σημείο που λέει ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η κυβέρνηση της χώρας κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της. Και παραλαμβάνω αυτά τα οποία είπε ο επικεφαλής του κ. Ιωραμπίδη, τα είπε ξεκάθαρα. Το τι γίνεται και τι γίνεται από κοινού. Και πώς χειριστήρια προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Βεβαίως υπάρχουν μεγάλα προβλήματα Πολλά από τα προβλήματα έχουν τις ρίζες τους στις ιστορικές αδικίες, αλλά με δεδομένο μας το Σύνταγμα, όπως λέει η έκθεση, προσπαθούμε να διορθώσουμε τα κακοσκήμενα. Να δούμε τι θα γίνει και σε εκείνο το κομμάτι της ε, χώρας του Το 80% της Κένιας είναι, είναι, είναι έρημο, είναι, ε, ε, είναι χέρσο. Το 80%. Το 20% πρέπει να θρέψει όλο τον πληθυσμό. Μιλούμε για 40 εκατομμύρια. Επίσης κάτι άλλο. Θα πρέπει να συνεργαστούμε. Να συνεργαστούμε και έτσι να πάμε σε κάποια βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, πιέζει ο χρόνο, οπότε παρακαλώ θέλω να αναγνωρίσετε ότι η ανθρωπιστική κρίση στην Κένια εν, εν μέρη οφείλεται σε αυτά τα οποία λέει η έκθεση, αλλά και από τις συγκρούσεις στην περιοχή και συγκεκριμένα από τις συγκρούσεις στην Σομαλία. Όλα αυτά μαζί ευθύνονται και άρα θα πρέπει έτσι να δείτε τα αποτελέσματα της διάσκεψης την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, είναι κάτι το οποίο φρενάρει πάρα πολύ τις αντισιακές προσπάθειες. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας. Η έκθεση είναι πάρα πολύ καλά τεκμηριωμένη. Σας ευχαριστώ και για τα συμπεράσματα που μας ε, δείχνουν ποιες είναι οι λύσεις. Ευχαριστώ. Σημειώνουμε τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Την παρουσία σας εδώ, τη δουλειά που έκαναν οι συγγητές, η προσωπία, την Επιτροπή για την παρουσία της, τον πρεσβευτή. Σας ευχαριστώ διάφορα. Ουχή. Ε, τότε λοιπόν, προσεχή συνεδρία 27 Μαρτίου, 12.30 με 3, 23 Απριλίου και 24 Απριλίου. Α, ναι, και να εφόσον και τους ερμηνείς που ξεπέρασαν ε, για άλλη μια φορά τα ε, ωράρια εργασίας.